Bonjour, cher collègue. On doit commencer. Καλημέρα συνάδελφοι, ξεκινάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Καλωσορίζω κυρίως τα μέλη των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών και φυσικά τα μέλη της Επιτροπής μας. Ανάμεσά μας έχουμε 36 βουλευτές από τα κοινοβούλια των κρατών μελών, 9 προέδρους και 3 αντιπροέδρους των αρμοδίων επιτροπών από 16 χώρες μέλη της Ένωσης και από 2 υποψήφιες χώρες, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία. Έχουμε επίσης και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από την Ορβηγία και την Ελβετία. Θεωρώ ότι το θέμα των συζητήσεών μας ε, σήμερα και αύριο, τα ευφυή e σύνορα, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, ε, ιδιαίτερα όταν η συζήτηση γίνεται ανάμεσα σε ευρωβουλευτές και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων. Είναι ευρωπαϊκό το θέμα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές καταστάσεις και πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί επηρεάζουν όχι μόνο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, χρησιμοποιήστε στο μέγιστο και στην αίθουσα αυτή, αλλά και κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λατκόφσκης, εξ ονόματος της Λετωνικής Βουλής. Έχετε το λόγο κύριε Λατκόφσκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου σε εσά για την πρόσκλησή σας, προκειμένου να συζητήσουμε τις εθνικές εμπειρίες όσον αφορά τη διαχείριση συνόρων και τις ευρωπαϊκές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το πακέτο αυτό ΕΦΗ σύνορα. Οι χώρες μέλη που μπήκαν στο Σέγγεν έπρεπε να αναλάβουν να συμμορφωθούν με τις κατάλληλες υποδομές και τον έλεγχο στα εθνικά τους σύνορα. Από τότε έχουν υπάρξει αρκετές αλλαγές έχουν εφαρμοστεί πολλά μέτρα για να ενισχυθεί ο έλεγχο στα σύνορα και η διαχείριση των σύνορων να γίνει πιο αποτελεσματική. Σήμερα οι χώρε μέλη αντιμετωπίζουν πολλέ προκλήσει που έχουν να κάνουν με διαχείριση σύνορων και δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα τη ασφάλεια, αλλά έχει να κάνει και με το θέμα τη διασφάλισης, των ρυθμίσεων, των σημείων ελέγχου, τη αποτελεσματικότητα, αλλά και την προστασία του ίδιου του προσωπικού ελέγχου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι δεν πρόκειται μόνο για τα αεροδρόμια, γιατί υπάρχουν και τα χερσαία σύνορα και τα θαλάσσια σύνορα. Με τι εξελίξει όσον αφορά τι επιχειρήσεις, την διακίνηση των ατόμων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και δεν σφάλουμε αν πούμε ότι όλοι μας έχουμε περάσει κάποιες ώρες μερικές φορές προκειμένου να περάσουμε τα σύνορα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου λοιπόν μας λέει ότι οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να βελτιωθούν, οι μηχανισμοί δηλαδή που διαθέτουμε να βελτιωθούν, αλλά συγχρόνως να προσέξουμε και ποιος θα μπορούσε να αποτελέσει η απειλή για παράνομη μετανάστευση. Η Λετωνία στηρίζει λοιπόν την χρήση των τεχνολογιών εχμής για αυτό το σκοπό τα η σύνορα, η πρωτοβουλία αυτή είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα. Και το προτινόμενο σύστημα εισόδου-εξόδου δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τους ελέγχους στα σύνορα και να χρησιμοποιήσουμε και ηλεκτρονικά μέσα για να ξέρουμε πόσο χρόνο μένει κανείς στις χώρες μας. Συγχρόνως το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών μας επιτρέπει πιο απλοποιημένες διαδικασίες στα σύνορα. Βεβαίω, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα του πειραματικού, του δοκιμαστικού αυτού προγράμματο ΕΦΗ e σύνορα, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την χρήση των διαδικασιών, των βιομετρικών στοιχείων και άλλων τεχνικών λύσεων. Όσο όμω συνεχίζεται αυτό το δοκιμαστικό πρόγραμμα, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσουν να συζητούν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ε, με θέματα που πάνε και πέρα από το πεδίο εφαρμογή του δοκιμαστικού αυτού προγράμματο. Πιστεύω ότι αναπτύσσοντας ένα νέο σύστημα εσόδου-εξόδου πρέπει να βασιζόμαστε σε ευρεία συστήματα πληροφοριών και να λάβουμε υπόψη μας επίσης και το κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν συμβατό με τα συστήματα που ισχύουν στις χώρες μέλη. Η εμπειρία μας δείχνει ότι χρειάζεται και ένα εθνικό σύστημα εισόδου-εξόδου. Είναι αποτελεσματικό αυτό και ανταποκρίνεται και στις ανάγκες όχι μόνο του ελέγχου στα σύνορα αλλά και της επιβολής του νόμου. Όσο προχωράμε λοιπόν με τα σύνορα, θυμίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει πάντα μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε απλοποίηση των διαδικασιών στα σύνορα, αλλά και της προστασίας των δεδομένων. Ειλικρινά πιστεύω και ελπίζω ότι η συνάντηση αυτή θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε επικοδομητικά τις προσπάθειές μας και θα προωθήσει το διάλογο ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λευκόφσκης. Τώρα Αρχίζουμε με το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας που έχει ως στόχο να μας επιτρέψει πραγματική πολιτική συζήτηση για τόσο διακυδεύονται με την πρόταση αυτή για τεφή σύνορα. Έχει υπάρξει μια τροποποίηση γιατί δυστυχώς ο κύριος Κοσλόφσκι δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας σήμερα για λόγους υγείας. Αντικαθίσταται από την κυρία Εβίκα Σιλινιά η οποία είναι υφυπουργό Εσωτερικών της Λετωνίας. Σας καλωσορίζω κυρία Σιλινιά. Είναι μεγάλη τιμή για μας βέβαια, γιατί έχουμε ανάμεσά μας και τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο, τον αναγνωρίσατε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους δύο εισηγητές μας, την Τάνια Φάγιον για το πρόγραμμα καταγραφής των ταξιδιωτών και τον κύριο Ντίας Ντεμέρα για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Θα ξεκινήσουμε με τους εισηγητές μας και στη συνέχεια θα, θα υπάρξει η ομιλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αυτοί που θα ήθελαν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης να το ζητήσουν το ταχύτερα δυνατόν για να καταλήξουμε σε ένα κατάλογο μιλητών. Για τον τρόπο τώρα που θα ζητήσετε το λόγο, θα ζητήσω από τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες που έχουν διάφορα χρώματα και είναι, ε, έχουν διανεμηθεί στην αίθουσα, είναι κίτρινα και ροζ. Κάθε χρώμα ανταποκρίνεται σε μία συνεδρίαση. Το κίτρινο αφορά την πρώτη, ε, το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης και το δεύτερο είναι ροζ. Καλείστε λοιπόν εφόσον θέλετε το λόγο για να θέσετε την ερώτησή σας να συμπληρώσετε αυτές τις αιτήσει. Οι κλητήρες θα τα μεταφέρουν εδώ. Για τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορείτε να σηκώνετε το χέρι σας ως συνήθως. Θα ξεκινήσουμε με δύο ερωτήσεις από εθνικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και μία ερώτηση εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο χρόνος ομιλίας θα είναι περιορισμένος σε σχέση με τον αριθμό πάντα των βουλευτών που θα ζητήσουν το λόγο. Οι κύριοι, κύριοι Φαγιόν και Μέρα θα έχουν τον λόγο για 15 λεπτά το πολύ που ξεκινάει τώρα. Η Τάνια Φαγιών λοιπόν έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω θερμά του συγκεκριμένου προσκεκλημένους μας, τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, την ε, Αναπληρώτρια Υπουργό, του συναδέλφου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων και όλους ιδιαίτερο όλους τους λοιπούς προσκεκλημένους και συμμετέχοντες. Ιδιαίτερη χαρά σήμερα η ευκαιρία που έχω να σας μιλήσω για το σημαντικό αυτό θέμα ως εισηγήτρια για το πακέτο των ευφύων συνόρων, των έξυπνων συνόρων Χαίρομαι που αυτή η σημαντική συνεδρίαση σήμερα λαμβάνει χώρα με την παρουσία όλων σας. Μια ακρόαση όπως η σημερινή νομίζω δείχνει ότι όπως πρέπει να συμβαίνει σε μια πραγματική ευρωπαϊκή οικονομία, η νόμη, η νομοθεσία που επεξεργαζόμαστε δεν φτιάχνεται για μας, αλλά για τους πολίτες μας. Έχουμε λοιπόν για άλλη μία φορά την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό και, σημαντικό και ευαίσθητο θέμα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που μας έχει απασχολήσει για χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που θα επηρεάσει σημαντικότατα τις θεμελιώδεις ελευθερίες για τους πολίτες μας στην Ευρώπη αλλά και την εικόνα έξω από τα σύνορά της που θα έχει η Ευρώπη, αλλά βέβαια και θα έχει και δημοσιονομικές συνέπειε. Αυτό που πάντα ακούγεται με την ακρόαση αυτή είναι τι κόστος θα συνεπιφέρει. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομία κλίμακος και τις διαφορετικές νομοθεσίες που υπάρχουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη, που θα πρέπει να αντικατασταθούν από μία που θα τις τροποποιεί, ήταν πολύ σημαντικό να συνομιλήσουμε, να συνδιαλεγούμε με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί από αυτά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του διαλόγου που θα αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο. Η δική σα δε εμπειρία, πρακτικέ που ενδεχομένω έχετε να προσφέρετε στην Τράπεζα των Συνομιλιών σήμερα, θα είναι πολύτιμα εργαλεία για τη δουλειά μα εδώ. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για την αθρώα προσέλευσή σα. Έχουμε εκπροσώπηση πολλών εθνικών κοινοβουλίων και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό σημάδι, μια σημαντική απόδειξη της ουσίας του θέματος. Είμαι λοιπόν συνεισηγήτρια. Με μεγάλη χαρά ε, συνεργάζομαι με τον Αγουστίν Διασδεμέρα Δεμέρα το θέμα αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε πραγματοποιήσει πολλές συζητήσεις, συναντήσεις με ειδικού, με σκιώδεις συζητητές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές τις δύο μέρες της συνάντησής μας θα ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εξελίξεις. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στο πρόγραμμα για το οποίο έχω αναλάβει εγώ την ε, τιμή της σύνταξης έκθεσης. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό θα έχει σαν ε, ουσία την διευκόλυνση της διέλευσης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων για τους ε, προερχομένους από τρίτες χώρες ταξιδιώτες κατά τρόπον που θα εξασφαλίζει ένα προκατακτικό έλεγχο πριν φτάνουν δηλαδή στο σημείο των συνόρων από μια πρώτη αντίληψη που έχω της κατάστασης, ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα πρέπει να δώσουμε, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε απαντήσει είναι εάν πράγματι σήμερα χρειαζόμαστε αυτά τα έξυπνα τα ευθύ σύνορα. Και ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της προτάσεως. Εάν ε, το προτινόμενο εγχείρημα έχει αναλογική ε, σχέση με το κόστος, με την επιβάρυνση, με την καθυστερήση. Εν τέλει, τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Ευρώπη φρούριο, όπου θα διώχνουμε τον ξένο ή μια Ευρώπη ανοιχτή, ανοιχτό χώρο με εγγύηση ελευθεριών και, πραγματικών, ε, και πραγματικά ελεύθερη διακίνηση. Αυτό το λέω διότι οι, οι δέσμοι μέτρων που έχουν κατατεθεί και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει και παράλληλα σε 12 κρατημέλη αφήνει πολλά ερωτηματικά ακόμη εκκρεμεί. Πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συζήτηση και με τον Επίτροπο που μας καθησύχασε λέγοντας ότι θα αναθεωρηθεί η νομοθετική πρόταση έως το τέλος του χρόνου και θα επαναυποβληθεί. Η αδιάκριτη λοιπόν συλλογή μαζικά δεδομένων χωρίς να υπάρχει επαρκής λόγος, από χρόνο λόγος, θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Και γι' αυτό θα πρέπει να διερωτηθούμε για την προστασία των συνόρων. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Ω προ το κόστο, ω προ την πρόσβαση των αρχών επιβολή του νόμου και ω προ τον όγκο των πληροφοριών, των δεδομένων που θα έλουμε να συλλέγεται. Περιμένω λοιπόν να ακούσω από εσά πώς βλέπετε το νομοθέτημα αυτό, ποια είναι η θεώρησή σας, ποιες είναι οι εθνικές εμπειρίες από ενδεχομένως αντίστοιχα συστήματα εθνικά. Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει σε 12 κράτη-μέλη πιλωτικά και σε 17 συνοριακά σημεία αεροπορικά, χερσαία και θαλάσσια. Ε, δοκιμαστικά, όπως είπα, ένα πρόγραμμα για την επαλήθευση του καλύτερου τρόπου διαχείρισης των δεδομένων αυτών. Άρα ανοιχτό παραμένει το ευαίσθητο αυτό θέμα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα για την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όπω ξέρετε έχει ήδη απορρίψει την προταθήσα νομοθεσία. Άρα, ποια είναι τα προβλήματα, σε ποια ερωτηματικά καλύτερα να δώσει απαντήσει η νομοθεσία, σε ποιο βαθμό προστατεύονται διαφορετικού τύπου σύνορα, τι απαντήσει μπορούν να δοθούν και σε ποιο βαθμό υφιστάμενα συστήματα που έχουμε, όπως το σύστημα πληροφοριών Schengen το ΒΙΣ, το Eurodac, σε ποιο βαθμό έχουν επιτύχει και σε ποιο βαθμό έχουν αποτύχει, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε τα εφιστάμενα πριν προχωρήσουμε στην εισαγωγή ενός νέου συστήματος. Επίσης, δε, οι προτάσεις που έχουμε, επιτάπητος και θα σας πει ο συνάδελφος Δεμέιρα περισσότερα για το συστημα εισόδων-εξόδων, εάν αυτά αναλογικά είναι τα κατάλληλα ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Αυτά είναι τα θέματα που θα μα απασχολήσουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι και εσείς και εμείς θα μπορούσαμε να βρούμε τις απαντήσεις αυτέ τι δύο μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριο Δία Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων όπως και από το Μαυροβούνιο, την Ελβετία και την ε, Νορβηγία. Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τη δουλειά σου που είναι πάντα πάρα πολύ πολύτιμη. Με 300.000 και παραπάνω σημεία στα σύνορα, με τόσους πολλούς πολίτες από τις χώρες μας που περνούν τα σύνορα, Προφανώς χρειαζόμαστε νέα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τις ροές αυτές. Και άλλοι δείκτες δείχνουν ότι τα σημερινά συστήματα πληροφόρησης, το sis 2 και το ΒΙΣ, δεν θα επαρκούν στο μέλλον προκειμένου να διαχειριστούμε μόνο με αυτά και από μόνο τους αυτά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ορών αυτών των 76 εκατομμυρίων επιβατών σε 302 σημεία διέλευσης το 2025. Υπό το φως λοιπόν των διαδικασιών ελευθέρωσης ή διευκόλυνσης των θεωρήσεων, σε κάθε περίπτωση βέβαια με ιδιαιτερότητες, έχουμε τα Βαλκάνια, έχουμε το Μαρόκο, έχουμε την Ρωσία. Όμως όλα αυτά μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε σοβαρά πώς θα εφαρμόσουμε τα ευφύ σύνορα. Είναι ένα νέο τοπίο, όπως είπε και η Τάνια πολύ σωστά. Αρχίσαμε από το 2008 με ανακοινώσεις, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ήθελε να εφαρμοστεί ένα σύστημα εισόδου-εξόδου. Από τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι η σημερινή διαχείριση των συνόρων μας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Διακυδεύονται πολλά συμφέροντα. Είναι λοιπόν δικιά μας υποχρέωση, αλλά και ευθύνη μας, να προχωρήσουμε με την πρόταση αυτή και να έχουμε μια νομοθετική απάντηση. Η ελευθερία διακίνησης είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να το διασφαλίσουμε, να το ενισχύσουμε το δικαίωμα αυτό και όχι να το αποδυναμώσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα τεχνολογικά στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε το σύστημα αυτό και το νομοθετικό αυτό πακέτο και η τρίτη έκθεση η οποία θα τροποποιήσει τον κώδικα Σέγγεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν τη διέλευση στα σύνορα των πολιτών μας και να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Λέμε πάντα παράτυπη εμείς, δεν λέμε παράνομη και να προλάβουμε και άλλα θέματα, άλλες απάτες, ε, ναρκωτικά, ε, λαθρεμπόριο κλπ. κλπ. Το θέμα των ε, διαβατηρίων, η καθυστέρηση όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την διαμονή, οι απάτες που γίνονται όσον αφορά την παραποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων. Είναι πράγματα που χρειάζονται λύση μέσα στο χώρο Σέγγεν. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε αξιόπιστα μέσα ώστε οι χώρες μέλη να μπορούν να καθορίσουν κατά πόσο κάποιος από μια άλλη χώρα έχει ξεπεράσει τον χρόνο παραμονής του ή όχι. Βασιζόμαστε στο άρθρο 77 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται εναρμόνιση λοιπόν κάποιων κανόνων που διαδιευκολύνουν τη διαχείριση και την χρήση της πληροφορίας που παίρνουμε από τις υπηρεσίες ελέγχου των συνόρων. Με εγγυήσεις βέβαια, πάντα με εγγύησει. Μία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την παράτυπη μετανάστευση ή τη διεθνή τρομοκρατία ή τα σοβαρά εγκλήματα. Τρεις χώρες μέλη διαθέτουν εθνικά συστήματα σήμερα που μοιάζουν αυτά τα οποία προτείνονται για το σύστημα εσόδου-εξόδου. Βέβαια διαφέρουν μεταξύ τους η πρόσβαση στο σύστημα, η διατήρηση των δεδομένων, ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται δεδομένα αυτά κλπ. κλπ. Οι διαφορές αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εσόδων-εξόδων, εσόδου-εξόδου μάλλον πιο σωστά, για να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Ξεκινούμε από την αρχή ότι χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα. Παρ' όλα αυτά πάρα πολλέ αμφιβολίες εκφράστηκαν. Το είπε και η Τάνια, πρόκειται για το θέμα το δημοσιονομικό, ότι ο στόχος δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος, η πρόσβαση στο σύστημα, η ασφάλεια κλπ. κλπ. Για όλου αυτούς τους λόγους λοιπόν και για να διευκρινιστεί περισσότερο η νομοθετική πρόταση, πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν αρχίσουμε με την τακτική νομοθετική διαδικασία, να περάσουμε από δύο στάδια. Το πρώτο θα ήταν μια τεχνική μελέτη, μελέτη αντικτύπου και δεύτερον να έχουμε ένα στάδιο συλλογής ε, στοιχείων. Έχουμε εδώ και τον ε, Διευθυντή της ε, Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αβραμόπουλε και εσάς που ήρθατε που είπατε τον Ιανουάριο του 2015 θα είχαμε μια νέα νομοθετική πρόταση αναθεωρημένη μία πρόταση στην οποία το 2016 πια θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την πρόταση αυτά και σήμερα είναι νομίζω ο κατάλληλος χώρος για να περάσουμε περισσότερο σε βάθος για την πρόταση αυτή. Χρειάζονται τεχνικά στοιχεία λοιπόν να περάσουμε από το δοκιμαστικό αυτό στάδιο για να καθορίσουμε την αρχιτεκτονική της νέας αυτής αναθεωρημένης πρότασης και να συζητήσουμε ό,τι περιλαμβάνεται στο νομοθετικό πακέτο. Εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή επίσης για να ζητήσω και διοργανικό διάλογο για θέματα τόσο σημαντικά όπως είναι η προστασία των δεδομένων. Θέμα πολύ βασικό για το Κοινοβούλιο μας, όπως επίσης η πρόσβαση στο σύστημα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή για το σύστημα που σφραγίζονται τα διαβατήρια. Βάσει λοιπόν του εγγράφου εργασίας θέλω να υποβάλω και κάποιο προβληματισμό σε σχέση με την συνάντηση αυτή. Σας είπα ότι πολύ με απασχολεί το θέμα των τεχνικών στοιχείων. Τι θα γίνει με τους επιτεχυντές επίσης της διαδικασίας. Θα έλεγα ότι κάθε μέτρο που εφαρμόζεται πρέπει να έχει όσο γίνεται μικρότερο αντίκτυπο στον ταξιδιώτη όσον αφορά το χρόνο, για παράδειγμα, που χρειάζεται για να περάσει τα σύνορα ή όσον αφορά τον περιορισμό των ε, ελευθεριών του δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία, όπως λέει και η τεχνική μελέτη. Να αφαιρέσουμε 10 από τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται μέχρι τώρα και να χρησιμοποιείται η διαδικασία με τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο στοιχεία που ήδη έχουν συλληφθεί. και να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα στοιχεία, το API, το VIS κτλ. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στα συμπεράσματα της ε, προσωρινής έκθεσης που μιλάει για αναλογικό ε, αριθμό στοιχείων που θα συλλέγονται, να κατοχυρωθούν δηλαδή αρχές αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Να υπάρχει επίσης και το θέμα της αναγνώρισης της ήρδας του ματιού ή του προσώπου. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στο νομοθετικό αυτό μέτρο, μην ξεχνάμε ποτέ τον στόχο μας. Να βελτιώσουμε τη διαχείριση των συνόρων δηλαδή, να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση, να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά είναι όμως θέματα που μας προβληματίζουν, που τα θέτω σε εσά στο σώμα. Γιατί η ελευθερία είναι πολύ βασικό στοιχείο για μας και από εκεί θα κρυθούν και το ποια στοιχεία χρειάζονται για να ολοκληρώσουμε το σύστημα αυτοδιαχείρισης των συνέρων που έχει να κάνει με τη ε, διατήρηση των δεδομένων, πόσο καιρό, ποιο θα έχει πρόσβαση κλπ. Τη θέση μου τη γνωρίζουν οι συνάδελφοι και αντιλαμβάνομαι ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί με τέτοια νέα συστήματα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητές τους. Υπάρχουν τα τεχνικά δεδομένα κύριος στόχος μας είναι η διαχείριση των ταξιδιωτών και η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά δευτεροβόντως πρέπει να δούμε υπό ποιε συνθήκε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και αρχέ επιβολή του νόμου για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία. Επ' αυτού βέβαια θα συζητήσουμε περισσότερο αύριο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ήθελα ευθύ από τώρα να σας γνωστοποιήσω τη δικιά μου τη θέση. Ένα άλλο θέμα εμβληματικό για μας είναι πώς θα συλλέγονται και πώς θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία. Δεν θέλω εδώ να μιλήσω για πολύ, αλλά πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Από το ΣΥΣ2, για παράδειγμα, Κάρλος, έτσι. Και να μην ξανακάνουμε τα ίδια σφάλματα που έχουμε κάνει και τα το παρελθόν. Ω Δημοσιονομική Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσέξει πάρα πολύ και όλα όσα έχουν να κάνουν με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο νέων μέτρων. Πρέπει να χρησιμοποιείται όσο γίνεται καλύτερα ο κοινοτικό προπολογισμό. Όλο ιδιαίτερο από πλευρά τη τεχνική αρχιτεκτονική πρέπει να μελετήσουμε τι είναι προτιμότερο. Ένα ενιαίο σύστημα και κατοχύρωση ταξιδιωτών και εισόδου-εξόδου ή δύο χωριστά συστήματα όντως είναι διαφορετικό το κόστος. Και πρέπει να αποφασίσουμε αν προτιμούμε αυτά τα δύο να είναι χωριστά ή ενιαία και αν πρέπει να συνδέονται με το ΒΙΣ ή όχι. Πρέπει ορθολογικά επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα τα οποία ήδη διαθέτουν οι χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα βελτιωθεί η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και θα αποφύγουμε επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τις επιπτώσεις της χρήσης όλων αυτών των συστημάτων μέσα στο χρόνο. Ειλικρινά, αυτό που προτιμάω είναι τον καλύτερο δυνατόν συντονισμό μεταξύ όλων των διαφορεμένων πλευρών, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική και πλήρη διαχείριση των συνόρων σημασία έχει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα το δημοσιονομικό του, κόστους δηλαδή. Πρέπει να ξέρουμε επακριβώς τι θα κοστίσει. Τέλος, το πακέτο αυτό, το νομοθετικό, πρέπει να πω ότι είναι πολύ φιλόδοξο. Και μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες αλλαγές. Τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά που πρέπει να αναλύσουμε είναι περίπλοκα. Οπότε ζητώ και εγώ, όπως έκανε και η συναδελφός μου η κυρία Φαγιόν, από όλες τις πλευρές που βρίσκονται εδώ σήμερα, να μας βοηθήσουν με τις δικές τους γνώσεις και πληροφορίες να βελτιώσουμε την νομοθετική μας αυτή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ντιμέρα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σιλινιά η οποία είναι η υφυπουργό εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λετωνίας. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάντηση αυτή αποτελεί προτεραιότητα της Λετωνικής Προεδρίας αποδεικνύει ότι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τις συζητήσεις, αλλά ελπίζω να δοθούν απαντήσεις στα ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και να διευκολύνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στα πλαίσια του προγράμματος καταγραφής των ταξιδιωτών. Έχουν γίνει πολλές επαφές ήδη ανάμεσα στο Συμβούλιο, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη του λεγόμενου πακέτου των εφιών συνόρων. Είναι ένα σημαντικό ε, τμήμα της προσπάθειας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να υπάρξει διευκόλυνση στις μετακινήσεις των πολιτών που επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν το πακέτο αυτό να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν και να γίνει αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα μειώσουμε τους χρόνους οι οποίοι απαιτούνται σήμερα και στα πλαίσια του ελέγχου των αιτήσεων και στα πλαίσια του περάσματος των συνόρων. Γνωρίζουμε ότι η χρήση των νέων ευκαιριών που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες δεν θα υπάρξει αν δεν υπάρχει ταυτόχρονο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμός των απορρίτων των προσωπικών. Επίσης η αύξηση του αριθμού των φυλάκων και ελεγκτών είναι κάτι το οποίο τίθεται. Δεν μπορεί κανείς μόνο να αφαιθεί αποκλειστικά στα ηλεκτρονικά μέσα. Πάντως μπορούμε και με το δεύτερο αυτό πρόγραμμα ελέγχου εισόδου και εξόδου ε, θα διευκολύνει ακριβώς ε, την καταγραφή των μετακινήσεων αυτών και θα μπορέσουμε για τον συγκεκριμένο ε, επισκέπτη να ορίζουμε σωστά και να ελέγχουμε σωστά τον χρόνο παραμονής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ξέρετε ότι κάτι τέτοιο με το σύστημα της φράγησης απλά των ταξιδιωτικών εγγράφων είναι ιδιαίτερος δύσκολο. Είναι επίσης σημαντικό να δίδουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες προς τους ταξιδιώτες σχετικά με την δυνατότητα παραμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος στα σύνορα θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, διευκολύνοντας τους επισκέπτες και επιτρέποντας να ανοιχνεύουμε ταχύτατα αυτούς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει ε, τον ε, χρόνο παραμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πακέτο αυτό ελπίζω ότι θα βελτιώσει την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και θα βελτιώσει επίσης και τους ελέγχους για λόγους ασφαλείας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο συμφέρει και τις τελωνιακές αρχές ή μάλλον καλύτερα τις ελεγκτικές αρχές γενικότερα στα σύνορα αλλά και τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Οι προτάσεις ε, που περιλαμβάνονται στο πακέτο δίδουν απαντήσεις σε τεχνικά προβλήματα και σε σχέση με το πρόγραμμα τακτικών ε, ταξιδιωτών και σε σχέση με το πρόγραμμα εισόδου-εξόδου. Η Προεδρία λοιπόν υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αρμόδιας Εξωτερικής Υπηρεσίας. Είμαι θα ευγνώμονες στα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τα πιλωτικά προγράμματα ε, στις μεθοριακές τους διαβάσεις. Υπάρχει όμως ακόμα μεγάλη ανάγκη να δοθούν απαντήσεις σε προβλήματα όπως η επιτάχυνση ε, των ε, διαδικασιών και η χρήση των βιομετρικών. Να υπενθυμίσω ότι η Ιταλική Προεδρία έχει ε, διασφαλίσει το ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ληφθεί υπόψη. Αυτό περιλαμβάνεται και στα συμπεράσματα του Κορεπέρ τον προηγούμενο Οκτώβριο. Οι εθνικές αρχές και η αρχή εποπτείας των προσωπικών δεδομένων θα εμπλακούν στην επεξεργασία των προγραμμάτων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν εμείς εκμεταλλευόμενοι ε, και την εμπειρία που έχουν οι μηχανισμοί ελέγχου και τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε να καταλήξουμε σε ένα σωστότερο πρόγραμμα. Θα συνεχίσει η Λετωνική Προεδρία λοιπόν ε, να ασχολείται με τα θέματα τα οποία τίθενται στη μελέτη και τα οποία δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστούν στο πιλωτικό πρόγραμμα. Θέματα τα οποία αφορούν τις ε, ε, συνέπειες της ανυπαρξίας δυνατότητας παρακολούθησης των κινήσεων των ταξιδιωτών, των διαφορών των διαδικασιών που ακολουθούνται σε διάφορες χώρες, και των διαδικασιών που αφορούν την καταγραφή των ταξιδιωτών στο πρόγραμμα των τακτικών κινήσεων. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε λοιπόν τα κράτη τα οποία έχουν ε, δώσει την υποστήριξή τους. Είναι επίσης ότι η πρόσβαση ε, των, των αρχών ασφαλείας στα στοιχεία αυτά δεν είναι ο βασικός στόχος. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλλά θα πρέπει να εκπληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν εθνικά συστήματα σε 13 χώρες που επιτρέπουν ε, την χρήση των στοιχείων που συλλέγονται στους μεθοριακούς σταθμούς. Ε, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αμοιβαία ενημέρωση και δεν υπάρχει και σωστός συντονισμός στα πλαίσια της χρήσης των στοιχείων αυτών και δεν υπάρχει δυνατότητα να συγκρίνουμε τα, τα στοιχεία που αφορούν την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την εμπειρία την οποία έχουν συλλέξει τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα. Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την αποτελεσματικότητα των νέων συστημάτων τα οποία θέλουμε να θέσουμε σε λειτουργία. Στην ομιλία του στις 21 Ιανουαρίου ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας μου είπε ότι η Λετωνική Προεδρία θέλει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του χρόνου Προεδρίας μας θα είμαστε σε τακτική βάση, σε επαφή μαζί σας και ελπίζουμε να βρούμε λύσεις και στα πολιτικά θέματα και επίσης και σε τεχνικά θέματα που αφορούν το πακέτο για τα ΕΦΗ σύνορα. Είναι απαραίτητο επίσης ε, να εξετάσουμε και την πρόταση του κυρίου Μωράες ε, για τον χρονισμό των επομένων συναντήσεών μας. Ευχαριστώ κυρία Σιλίνια. Αγαπητοί συνάδελφοι των, Ευρωπαϊ... των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να συμπληρώνετε το κίτρινο φυλάδιο, το κίτρινο έντυπο, προκειμένου να λάβετε μέρος στις συζητήσεις. Εν τω μεταξύ δίνω το λόγο όμω στον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης εσωτερικών και ηθαγένειας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Λιάννα αξιότιμα βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχά, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να συζητήσω και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ε, ιδέες για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι τα ΕΦΗ σύνορα και την ανάγκη για τον εξυγχρονισμό τον, ε, του τρόπου διαχείρισης των ευρωπαϊκών σύνορων. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε λεπτομερώς αυτή την πρόκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την το Προεδρείο και την Γραμματεία της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία αυτή, την Λετωνική Προεδρία και τους εισηγητές, την κυρία Φαϊόν και τον κύριο Διαστεμέρα για την προσήλωσή τους και τη δουλειά τους σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Οι σημερινέ παρουσιάσει δείχνουν για άλλη μια φορά ότι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει κρίσιμη σημασία για τις κοινέ προσπάθειές μας, Θα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εφιών συνόρων που θα ανταποκρίνεται στους στόχους του και θα προσφέρει αποτέλεσμα ανάλογο με το μέγεθος της πρόκλησης και της δαπάνης. Όπως αναφέρθηκε, νωρίτερα. Βρισκόμαστε σε μια φάση μεταξύ δύο νομοθετικών προτάσεων. Αλλά πιστεύω ότι αυτή την περίοδο μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να εμβαθύνουμε στον ε, διάλογο και να ανταλλάξουμε απόψεις με τρόπο ειλικρινή. Η αρχική πρόταση, νομοθετική πρόταση για τα εφικά, εφή σύνορα, είχε κάποια ζητήματα, τόσο τεχνικού όσο και πολιτικού χαρακτήρα, αλλά και οικονομικού σχέση με το κόστος που θα συνεπέφεραν. Αυτά τα επισήμαναν τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο. Όπως ήδη ανακοίνωσα, η δοκιμαστική περίοδος, τόσο με την τεχνική μελέτη, όσο και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης, μαζί με τα αποτελέσματα των συζητήσεων με εσάς, με το Συμβούλιο και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, θα αποτελέσουν την ε, τροφή για τη νέα πρόταση, νέα νομοθετική πρόταση που πιστεύω ότι θα, είναι, θα σε θέση να καταθέσουμε στις αρχές του 2016. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταθέτοντας τη νέα νομοθετική πρόταση, θα αποσύρει τις προτάσεις του 2013. Αναφέροντας λοιπόν τις προτάσεις μας, θα πρέπει να κοιτάξουμε για άλλη μια φορά τα ευρύτερα ερωτηματικά που γεννώνται άλλωστε και από τη σημερινή συζήτηση. Πρώτον, γιατί χρειαζόμαστε ευφυή σύνορα. Δεύτερον, τι επιδιώκουμε με αυτά. Και τρίτον, αξίζει το κόστος που συνεπιφέρουν αυτά τα νέα συστήματα. Η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα είναι ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη διαχείριση των ροών ταξιδιωτών τα κράτη-μέλη και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων προκύπτουν από τον κώδικα συνόρων του Σέγγεν. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει σε περίπτωση διαχείρισης διαλέψεως υπηκών τρίτων κρατών, διότι τότε καλούνται να επαληθεύσουν την ε, γνησιότητα και εγκυρότητα των ταξιωτικών εγγράφων, την κατοχή όπου χρειάζεται έγκυρης θεώρησης διαβατηρίου, τον στόχο και τους όρους της διαμονής και την πιθανή ύπαρξη σήματος από το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, τα κράτη. Έχουμε λοιπόν ε, με βάση εκτιμήσεις μας περίπου 200 εκατομμύρια διελεύσεις συνόρων από υπηκόους τρίτων κρατών κατά την είσοδο ή την έξοδο από το χώρο Σέγγεν. Και θεωρούμε ότι στην προσεχή δεκαετία θα αυξηθεί αυτός ο όγκος κατά ακόμη 100 εκατομμύρια διελεύσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με σημαντική επιβάρυνση σε υποδομές και ανθρώπινους πόρους στα εξωτερικά μας σύνορα. Το ζήτημα δεν είναι βέβαια μόνο να αντιδράσουμε σε αριθμητικά στοιχεία, να διαχειριστούμε νούμερα. Έχει να κάνει όλη αυτή η προσπάθεια και με την ποιότητα των ελέγχων στα σύνορα. Με το υφιστάμενο σύστημα τα, οι 200 εκατομμύρια διελεύσεις των συνόρων συνεπάγονται ότι 200 εκατομμύρια φορές ένας υπάλληλο, ένας συνοριοφύλακας, χτυπάει τη σφραγίδα του πάνω στο διαβατήριο ενός ταξιδιώτη. Οι συνοριοφύλακες σήμερα κάνουν ε, έλεγχο μη αυτοματοποιημένο στα ταξιδιωτικά έγγραφα, επαληθεύουν δηλαδή τις ημερομηνίες εισόδου-εξόδου, υπολογίζουν τη διάρκεια διαμονής. Πολλές φορές το, η δυσκολία έγκυται στο ότι είναι δυσανάγνωστη σφραγίδα και πάντως όλες αυτές τις πληροφορίες δεν καταχωρίζονται πουθενά. 12 λοιπόν κράτη Σέγγεν και Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ήδη εισαγάγει συστήματα εθνικά εισόδων-εξόδων και ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα του χώρου του Σέγγεν, αλλά ταυτόχρονα και ε, η Πορτογαλία και η Κύπρος, σημαίνουν 13 συστήματα εθνικά μη συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, εάν ένας ταξιδιώτης μπει στο χώρο Σέγγεν μέσω ενός από αυτά τα κρατημέλη, αλλά βγει από το χώρο Σέγγεν από ένα άλλο κράτος μέλος, δεν υπάρχει αντιστοίχηση των πληροφοριών μεταξύ των δύο συστημάτων. Επίσης υπάρχουν ε, αποκλήσεις μεταξύ των συστημάτων, των εθνικών αυτών συστημάτων, επί παραδείγματι ως προς το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται ή τη διάρκεια της διακράτησής τους. Το εφιστάμενο λοιπόν σύστημα ούτε αποτελεσματικό είναι, ούτε εξυπηρετεί το στόχο του όπως θα έπρεπε. Και άρα η αδράνεια δεν είναι η σωστή λύση. Πρέπει να βελτιωθούν τα σύνορα και με τη χρήση της τεχνολογίας πρέπει να καταστούν πιο ευφύοι, πιο έξυπνα. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε και πιο πολύ ώρα αναμονή στα σύνορα και ενδεχομένως απασχόληση περισσότερων ή και απασχόληση περισσότερων συνοριοφυλάκων, πράγμα το οποίο δεν είναι αποδεκτό ή εφικτό. Το σύστημα των ευφυών συνόρων με την ε, συστηματική λοιπόν καταγραφή όλων των εισερχομένων και εξερχομένων υπηκών τρίτων κρατών, αυτοματοποιημένο, θα μπορέσει να ελαχιστοποιήσει το χρόνο διέλευση από τα σύνορα. Και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η περίοδος δοκιμής, επαλήθευσή του. Με την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ευφυών σύνορων του Σέγγεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκομίσει πολύ περισσότερα ωφέλη από όσο θα χρειαστεί να κοστίσει η εισαγωγή του συστήματος και οπωσδήποτε πολύ προσθέτω πόσο δαπανούν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη χωριστά στη διαχείριση των σύνορων τους. Αντί λοιπόν να χρειαστεί να ε, απασχολήσει περισσότερο συνοριοφύλακες το κάθε κράτος μέλος, θα μπορούσε να ενισχύσει τη στελέχωση άλλων υπηρεσιών που, παραδείγματι, θα είχαν να κάνουν με τη μετανάστευση και δι' το άσυλο. Ε, ο δε κύριος στόχος ε, του συστήματος διαχείρισης συνόρων Σέγγεν θα ήταν η προαγωγή της κινητικότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ, Ευρωπαϊκή, ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Άρα θα σήμαινε αυτό επιτάχυνση και διευκόλυνση των διελεύσεων για τους τακτικούς ταξιδιώτες. Επίσης θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η, αποτελεσματικός ο εντοπισμός εκείνων οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους της διαμονής τους στην, ε, στον χώρο του Σέγγεν, θα μπορούσαν τα ευφύ αυτά σύνορα εκ τούτου να συμβάλλουν σε μια ασφαλή μεν, ανοιχτή δε Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα καλωσορίζει και τον τουρίστα, τον επιχειρηματία και οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη και θα αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για όλους. Θα επέτρεπαν επίση ώρα την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων. ενοποιημένα δεδομένα για εκείνους που ε, ξεπερνούν τα όρια της διαμονής τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα, ε, χρήσιμες πληροφορίες για ε, ενδεχόμενη αναθεώρηση μελλοντικών πολιτικών για τη μετανάστευση. Παραδείγματι, θα μπορούσε να εντοπιστεί από το σύστημα εισόδων-εξόδων ότι κάποιοι υπήκοοι συγκεκριμένη προελεύσεω, συγκεκριμένου κράτου δηλαδή, τρίτου κράτου, τείνουν να ξεπερνούν τα όρια της διαμονής τους, τα όρια της θεώρησής τους. Και αυτό θα μπορούσε να είχε σαν συνέπεια την ε, εισαγωγή μιας υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίων για την εν λόγω χώρα ή και την άρση, εάν συνέβαινε το αντίθετο. Επίσης αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και για τις ε, πολιτικές ε, επανεισδοχής. Θα ήθελα λοιπόν, ολοκληρώνοντας, να επισημάνω ότι η απόφαση μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί. Έχουμε, ακόμα αξιολογούμε όλα τα επιχειρήματα που προβάλλονται. και ιδιαίτερα θα μας απασχολήσει το ζήτημα της πρόσβασης για τις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για να ακούσω προσεκτικά όλα τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται. Περιμένω να συνεχιστεί αυτή η ανταλλαγή απόψεων για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Η αξιολόγηση συνεπειών του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα που παράγονται από το σύστημα εισόδων-εξόδων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις αρχές για την επιβολή του νόμου ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και λοιπόν σημαντικών αδικημάτων, ποινικών αδικημάτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για εντοπισμό ε, υπετίων και ως ένα εργαλείο διάγνωσης των εγκλημάτων, εγκληματολογικού τύπου. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ούτε για την αναγκαιότητα, ούτε για την αναλογικότητα της χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα εισόδων-εξόδων του, ε, για τις αρχές επιβολής του νόμου. Μια ενδελεχής λοιπόν αξιολόγηση χρειάζεται και με βάση τα όσα ορίζει η οδηγία για την διακράτηση προσωπικών δεδομένων. Εφόσον χορηγηθεί όμως η πρόσβαση στις αρχές επιβολής του νόμου, η απαραίτητη, ουσιαστική, ε, θα χρειαστεί να εισαχθούν τα απαραίτητα, ε, οι απαραίτητες ουσιαστικές και δικονομικές δικλίδες ασφαλείας, όπως ορίζει και το δικαστήριο στην ομολογία του με την ε, παρουσίαση μου σήμερα επικεντρώθηκα στα ευρύτερα ζητήματα που καλύπτει αυτή η πρώτη σας συζήτηση κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολύ πιο λεπτομερή και πολύ σημαντικά επιστεχνικού χαρακτήρα ζητήματα που θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρία. Συζήτηση και μελέτη όλων αυτών των θεμάτων συνεχίζεται. Έχουμε να κάνουμε με την ε, ε, με τις συνέπειες της κατάργησης της φράγησης και ιδιαίτερα σε σχέση με τους ε, ε, κατόχους άδειας παραμονής και τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την μη διαθεσιμότητα του συστήματος. Θα χρειαστούν επιπλέον συζητήσει και συναντήσει τεχνικού τύπου μεταξύ Επιτροπή και Κοινωνία των Πολιτών, μεταξύ φορέων διαχείριση, μεταξύ υπηρεσιών που εξασφαλίζουν τις μαζικές μεταφορές, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τα κράτη-μέλη που έχουν τα εθνικά συστήματα, τρίτες χώρες που εμπλέκονται κτλ. Από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και ανταλλαγές απόψεων θα τροφοδοτηθεί η διατύπωση της νέας αξιολόγησης συνεπειών και οι νέε νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες όπως είπα ελπίζω να είμαστε θέση να δούμε στον πρώτο μήνα του 2016. Η σημερινή συνεδρία είναι ένα πολύ σημαντικό ε, βήμα σε αυτή τη ε, διαδικασία συνεργασίας. Προσβλέπω και προγραμματίζω περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας. Πιθανώς δεν δε και μια κοινή ε, διερευνητική αποστολή σε συνεργασία με τους συνεισηγητές. Η δουλειά όμως έχει ξεκινήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή συνέχιση στη δουλειά σας καλύτερα στη δουλειά μας, στις εργασίες μας, σήμερα και αύριο. Και όπως είπα και στην αρχή, λυπούμε ιδιαίτερος που θα χρειαστεί να αποχωρήσω αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησή μου. Όμως ο διευθυντής μας που είναι πολύ κατηρτισμένος στα θέματα αυτά, γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες η διευθυντριά μας, κυρία Μπελίντα Πικ, είναι εδώ, θα σας δώσει λεπτομέρειες απαντήσει σε κάθε ερώτημά σα εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Είναι προφανέ ότι στη διαδικασία αυτή τη προετοιμασία των νέων προτάσεων θα έχουμε περισσότερε ευκαιρίε να συζητήσουμε μεταξύ μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και συνεργασία σας. Ευχαριστούμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Δύο ερωτήσει από τα Εθνικά Κοινοβούλια, μία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Σιμπάρες, προφέρω καλά το όνομα, αναρωτιέται πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων από τη Λιθουανία. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο πιο πολύ, όχι τόσο ερώτηση. Η Λιθουανία πρώτα απ' όλα είναι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της όσον αφορά το πακέτο ΕΦΗ σύνορα. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι το πρόβλημα μας είναι γνωστό. Η Λιθωνία από την αρχή στήριξε την πρωτοβουλία αυτή. Είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι η χρήση εφιών τεχνολογιών και εφιών ελέγχων στα σύνορα είναι κάτι αναπόφευκτο. Διότι θέλουμε να έχουμε από τη μια μεριά υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου στα σύνορα, από την άλλη μεριά θέλουμε να διασφαλίσουμε φιλικούς προς τον ταξιδιώτη ελέγχο στα σύνορα. Έχουμε όλο και περισσότερους ταξιδιώτες που περνούν τα σύνορά μας. Οπότε μόνο με τέτοια ευφύ σύνορα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις που τίθεται. Μόνο έτσι, εξάλλου, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Έχουμε ένα σύνορα με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και έχουμε και προς το Καλίνιγκρατ έναν διάδρομο transit. Η Λιθουανία λοιπόν είναι από τις 13 χώρες μέλη που έχουν το δικό τους σύστημα εισόδου-εξόδου. Ένα σύστημα πολύτιμο πραγματικά, αλλά όπως πολύ σωστά είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στην ζώνη Σέγγεν, και εμείς συμμετέχουμε στο σύστημα Σέγγεν, οι ταξιδιώτες μπαίνουν από μία χώρα, αλλά μπορεί να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από μία άλλη χώρα. Γι' αυτό και πρέπει να συνδυάζονται τα συστήματα αυτά. Και συμφωνώ και με την Υπουργό της ε, Λετωνίας που είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το σύστημα αυτό για όλα τα σύνορα, και τα χερσαία δηλαδή, και τα θαλάσσια και τα ενέργεια. Τα τρία ευρωπαϊκά συστήματα πάντως σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στον μελλοντικό τους ρόλο. Γιατί όταν φτιάχτηκαν η ιδέα ήταν εντελώ διαφορετική. Και πιστεύουμε ότι η συμβατότητα των ε, υπαρχών των συστημάτων με τα νέα που προτείνονται είναι κάτι αναγκαίο. Άρα πρέπει να δούμε και την υπόθεση του κόστους. Συνεπώς είμαστε υπέρ της εισαγωγής και του συστήματος εισόδων εξόδων και του συστήματος καταχώρησης ταξιδιωτών. Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν πάντως και περιμένουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περίοδου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ερώτηση. Από την κυρία Κατηρίκλη Ελβετία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Ρικλίν. Ναι. Είμαστε από την Ελβετία μέσα στο σύστημα Σέγγεν και είμαστε υπέρ της σημερινής πρότασης. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κύριος στόχος του συστήματος είναι μια αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Σέγγεν, ελέγχοντας τις εισόδους και τις εξόδους υπηκών χωρών. Όπως ήδη αναφέρεται στο, στην πρόταση εργασίας, ήδη από το 2014 αποφασίσαμε ότι υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης των αρχών επιβολής των νόμων που είναι ο ε, επόμενος στόχος του συστήματος. Η πρόσβαση αυτή όμως πρέπει να λάβει υπόψη την εμπειρία που έχουμε με τα μέχρι τώρα συστήματα, με το ΣΥΣ δηλαδή. Όπως είπαν και οι χρειάζεται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας που να διασφαλίζεται πάντα και για όλους. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο Ιγνάσιο Κάσης να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, η αναλογικότητα και η αναγκαιότητα, η αρχή αυτή δηλαδή, πρέπει να τηρείται και μέσω του συστήματος καταγραφής εισόδων-εξόδων και της καταχώρησης των ταξιδιωτών. Και όντως αναφέρονται οι αρχές αυτές. Για να λειτουργήσει καλά το σύστημα αυτό από την αρχή, η Ελβετία πιστεύει ότι τα βιομετρικά στοιχεία πρέπει να συλλέγονται από την αρχή ή τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τουλάχιστον την εικόνα του προσώπου. Όσον αφορά το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών, περιμένουμε τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περίοδου. Όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτά, θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε κατά πόσο τελικά θα στηρίξουμε μια τέτοια αναλλακτική πρόταση, όπου το σύστημα αυτό καταχώρησης ταξιδιωτών θα χρησιμοποιεί βιομετρικά ε, στοιχεία από το σύστημα ΙΕΣ e και Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι ξέρουμε, σκοπεύει τον Σεπτέμβριο φέτος να υποβάλει νέες προτάσεις. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σας της ΛΥΜΠΕ για την πρωτοβουλία αυτά, αυτή και τι λένε οι άλλες χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν ε, άκουσα το όνομά σας. Και τώρα, ο κύριος Κουαγιό. Είναι συναδελφός μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την ομάδα του ΕΛΚ, που εργάζεται πολύ πάνω στα θέματα Σέγγεν και διαχείρισης συνόρων. Παρακαλώ κύριε Κουαγιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, συμφωνώ με την ιδέα που ανέφεραν πολλοί ομιλητέ μέχρι τώρα, ότι δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώ η περιοχή Σέγγεν και η ελευθερία διακίνηση. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συνεργαστούμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί η αμοιβή εμπιστοσύνη είναι και το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαχείρισης των συνόρων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πολύ τους δύο εισηγητές μας, την Τάνια Φανιών και τον Αγκουστίν Διαθντεμέρα, για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, στόχος. Πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Ποιος είναι ο στόχος του συστήματος αυτού. Στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος ήταν να ελέγξουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. για να ελέγξουμε αυτούς οι οποίοι ξεπερνούν τον ε, χρόνο παραμονής για τον οποίο έχουν μια άδεια. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της ε, ευθυγράμμισης των νομοθεσιών μας. Συζητήσαμε λοιπόν για ένα αρμοσμένο σύστημα σχετικά με το οποίο δεν έχουμε κοινή πολιτική. Από την άλλη μεριά είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι θέλουμε να δούμε και ένα σύστημα που να μην ελέγχει μόνο το 25% των δουλεύσεων. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξή. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μα. Τα χρησιμοποιούμε καλά τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μα. Και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε ότι το SIS δεν χρησιμοποιείται ακόμα πλήρως. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της πλήρους αξιολόγησης της χρήσης των συστημάτων SIS και VIS. Και η τρίτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το κόστος. Όπως είπε και ο Κωστίν δεμέρα, πρέπει να μην ξεχνάμε τα μαθήματα που πήραμε από το SIS 2. Και το πρώτο είναι ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε ένα σύστημα το οποίο μας κόστησε 8 φορές παραπάνω από ό,τι είχαμε εκτιμήσει αρχικά. Πρέπει να είμαστε Ειλικρινεί λοιπόν όταν μιλάμε για κόστος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα κόστος και μετά να διαπιστώσουμε ότι μας στοιχίζει 8 ή 5 φορές ή έστω και 2 φορές παραπάνω από ό,τι αρχική εκτίμηση. Το είπε και η Τάνια Φαγιών αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια επίση πρέπει να συνεργαστούν. Γιατί στο τέλος πρέπει να αξιολογήσουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Και σε αυτήν την ερώτηση πρέπει να απαντήσουμε και θα τελειώσω με αυτό. Τα χρήματα τα οποία θα επενδύσουμε στο σύστημα δικαιολογούν τις πληροφορίες και το φέλη που θα πάρουμε από την εφαρμογή του συστήματος. Αυτή είναι μια βασική ερώτηση στην οποία καλούμε όλοι να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόγιο. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κρασκάλος, Πολωνία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι παρουσιάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό θα είναι απαραίτητο και χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας σκεφτούμε τις τελευταίες στατιστικές που έχουμε στη διάθεσή μας, θα δούμε ότι ο αριθμός των μη νομίμων μεταναστών ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες και να μην ξεχνάμε και αυτούς οι οποίοι ε, περιμένουν στα σύνορα. Θα πρέπει το σύστημα για να πετύχει να είναι αποτελεσματικό, ορθολογικό και απλό στη χρήση του. Και σε επίπεδο διαδικασίας φυσικά ε, για τους ταξιδιώτες. Πώς θα το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να συνδυάσουμε το σύστημα εισόδου-εξόδου με το σύστημα καταχώρησης. Πρέπει να συνδέσουμε τα δύο αυτά συστήματα δηλαδή. Απαιτείται αυτό να γίνει και στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και στα πλαίσια της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σύνορα αυτά. Δεν θα πρέπει το χειμώνα να αγοράζουμε μία Mercedes ε, και ε, το καλοκαίρι να ενθυμούμεθα ότι δεν αγοράσαμε σύστημα κλιματισμού. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε επίσης ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν εντελώς διαφορετικά συστήματα. Στην Πολωνία σαν παράδειγμα θα έπρεπε να είχαμε 60 επιπλέον ε, υπαλλήλους κάθε υπάλληλο κοστίζει σε αιτήσια βάση ένα κάποιο ποσό και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας με τον σωστότερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να υπάρξει επίσης σωστός τρόπος κατανομής του κόστους ανάμεσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το πρόβλημα με την ηλεκτρονική και την τεχνολογία είναι ότι μερικές φορές το σύστημα δεν θα δουλεύει. Τι θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση, έχετε προβλέψει κάποια λύση. Ο κύριος Οβίντιου από την Ρουμανική Γερουσία, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρουμανία ε, καλύπτει ένα τμήμα αρκετά σημαντικό των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολείται και με ένα μεγάλο κομμάτι της ασφάλειας των συνόρων του Σέγγεν. Υποστηρίζουμε φυσικά τα μέσα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και υποστηρίζουμε και τον καθορισμό αυτών των νέων συστημάτων ελέγχου που ονομάζουμε πακέτο εφιών συνόρων. Αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε κάποια πολιτικά κριτήρια τα οποία συχνά δεν είναι ορθά. Εμείς θέλουμε να αξιολογηθούμε με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να ενταχθούμε το ταχύτερο δυνατόν στη ζώνη Σέγγεν. Στην περίπτωση κατά την οποία βέβαια θέλουμε να πετύχουν αυτά τα ευφυή σύνορα. Ευχαριστώ κύριο Βιδίου. Κυρία Τσίπελ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την Επιτροπή Λίγκ Μπλίμπε, Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για την περαιτέρω συζήτηση να κάνω κάποιες ε, υποδείξεις αλλά να διατυπώσω και κάποιες ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι σε τι μας χρειάζεται το σύστημα. Σίγουρα δεν το χρειαζόμαστε δεδομένης της επιβάρυνσης για, και του κόστους για να μειώσουμε τις ουρές στα σύνορα. Δεν είναι αυτό επαρκής αιτιολόγηση. Για τον overstayer, αυτόν που ξεπερνάει δηλαδή τον χρόνο παραμονής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός ή τόσο μεγάλος κίνδυνος που προκύπτει από εκείνους που ξεπερνούν τη διάρκεια παραμονής της θεώρησής τους, ώστε να δικαιολογείται η επιβάρυνση. Από την άλλη πολύ συχνά λέγεται ότι με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων γίνονται πιο ασφαλή τα σύνορα. Μα τους τελευταίους ακριβώς μήνες ήρθαν πολλές ε, πληροφορίες από πρακτικές δοκιμές όπου και το σύστημα ακόμη του δακτυλικού αποτυπώματος μπορεί να παραποιηθεί αλλά και της αναγνώρισης προσώπου και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Ο κύριος Διασδεμέρα είπε ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα όπου μπορεί να μην είναι επαρκή για αποτελεσματικούς ελέγχους όπως το σύστημα SIS. Δεν θα ε, φέρω εγώ αντίρρηση, αλλά το ΣΥΣ και άλλα συστήματα που έχουμε δοκιμάσει δεν έχουν αξιοποιηθεί πολλές φορές σύμφωνα με το στόχο τους από τα κράτη-μέλη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν σε τι θα ωφελήσει να σχεδιάσουμε ένα νέο και δαπανηρό μέσον εάν τα κρατη δεν έχουν την πρόθεση ή δεν έχουν τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλά μέτρα για την ασφάλεια, πάνω από 200 μέχρι τώρα, που θα περιπλέξουν ακόμη τώρα την κατάσταση. Επίσης, Ποιος μπορεί να περνάει τόσο εύκολα τα σύνορα, τόσο γρήγορα. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος ταξιδεύει τακτικά ε, και λέει ότι θα παίρνει ηλεκτρονική σφραγίδα κτλ. Μα νομίζω ότι υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες είναι αυτοί που λένε ότι ένας επιχειρηματίας που έρχεται τακτικά χωρίς να δημιουργεί προβλήματα μπορεί να πάρει τη σφραγίδα του εύκολα χωρίς δυσκολίες. Αλλά ότι αντίθετα αυτός που δεν τηρεί τις προϋποθέσεις θα έχει προβλήματα. Τι γίνεται σε περίπτωση άρνησης της διέλευσης, ε, πώς θα διαπιστώνετε αν, κάποιος, αν σε κάποιον πρέπει να αρνηθούμε τη διέλευση και πού θα μπορέσει να προσφύγει αυτό σε περίπτωση που έχει απορριφθεί η δυνατότητα διέλευσης, εισόδου. Μια σειρά λοιπόν από παραμένουν ανοιχτά. Όπως επίσης η ποινική διαχείριση του ζητήματος. Κρίσιμα ζητήματα γιατί και η παράτυπη μετανάστευση και η υπόσταση ενός ποινικού αδικήματος βλέπω να μπαίνουν μαζί σαν θέματα προς διαχείριση. Και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω, παράτυπη είσοδος σημαίνει αυτομάτως ποινικό αδίκημα δεν θα πρέπει να προσδιοριστούν ε, ε, προϋποθέσεις. Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα, πώς πάνε σε κεντρικά συστήματα και πώς περαιτέρω διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα χρειαστεί να το μελετήσουμε για πολύ καιρό ακόμη. Ευχαριστώ πολύ Μπιρκίτ. Από τη Μάλτα τώρα ο συναδέλφος κύριος Ζάμιτ. Έχουμε ένα θέμα με τα μικρόφωνά μας προς το παρόν. Θα επανέλθουμε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορούμε να περιμένουμε δύο λεπτά μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα. Δεν έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε μαλτέζικα, δεν προβλεπόταν στην συνεδρίαση η μαλτέζικη γλώσσα. Αχ, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι προβλεπόταν. Θα μιλήσω αγγλικά όμω. Λυπούμε πολύ κύριε Ζάνιτ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν, το οποίο πράγματι ε, επηρεάζει και αφορά όλες μας τις αξίες. Ιδιαίτερα σε χώρα όπως η Μάλτα. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο μας επηρεάζει άμεσα μάλιστα γιατί είμαστε χώρα στα άκρα του Σέγγεν, παραμεθόριος, και άρα έχουμε να κάνουμε θέματα τα οποία επηρεάζουν τη χώρα μας ευθέως, αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για μας λοιπόν, εμείς έχουμε ένα σύστημα εθνικό εισόδων-εξόδων, όπου συλλέγονται ψηφιακά δεδομένα ταξιδιωτών, ένα σύστημα πολύ σημαντικό, εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας μας και διευκολύνει βεβαίως και τους ταξιδιώτες. Ε, για τα ζητήματα που έχουν εγερθεί σε σχέση με την αντιστήχηση των δεδομένων, όταν ε, παραδείγματι έχουμε είσοδο από τη, στη Μάλτα ενός του κράτους, ο οποίος όμως συνεχίζει μέσα στο Σέγγεν για να βγει από, την Ευρωπαϊ... από το χώρο Σέγγεν από άλλη χώρα μέλος, ή το αντίστροφο, η αντιστοίχηση αυτών των στοιχείων, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο Επίτροπος, αλλά έχει σημειωθεί και από άλλους ομιλητές, Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πλέον να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να διευκολυνθεί αυτή η αντιστοίχηση. Έχουμε όλο και περισσότερες διελεύσεις σύνορων, ακόμη και στο δικό μας επίπεδο το πιο περιορισμένο, και πρέπει επιτέλους να δούμε, ιδιαίτερα για να γίνει μια ε, ανοιχτή ε, περιοχή η Ευρώπη και όχι ένα φρούριο, να είναι ελκυστική δηλαδή προς ε, τον ταξιδιώτη, η οποία θα διευκολύνει αυτή την αντιστοίχηση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ε, οποιαδήποτε απόφαση να αναλάβουμε θα πρέπει να τη λάβουμε, πιστεύω, βάσει των αξιών και κυρίως του άρθρου 2 της συνθήκης. Σεβασμό δηλαδή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπων δικαιωμάτων. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με βάση αυτές τις αξίες. Αυτά τα λέω διότι η συλλογή, η διαβίβαση, η χρήση, η κοινή χρήση δεδομένων προσωπικών ενέχει και τον κίνδυνο της παραβίασης αυτών των βασικών αξιών και των θεμελιωδών ελευθεριών. Άρα θέλουμε οποιαδήποτε διαδικασία εισαχθεί να καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση από Εθνικό Κοινοβούλιο για τον κύριο Ντίντσερ, Τουρκικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής εδώ. Η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε μία πρόταση για τους υπηκόους τρίτων κρατών που θέλουν να, εισα... να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο Schengen σύστημα πληροφοριών Schengen και πρέπει αυτοί να καταγράφονται με βάση την νομοθεσία. Να καταχωρίζονται τα στοιχεία τους για μας μια τέτοια πρόταση δεν παρουσιάζει προβλήματα, θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Σε περίπτωση που γίνεται απλώς έλεγχος διαβατηρίων, διαχειρός όπως θα λέγαμε, ε, μπορεί να προκύψουν χρήσεις παραποιημένων ή πλαστών διαβατηρίων. Άρα χρειάζονται και τα βιομετρικά συστήματα οπωσδήποτε. Με ένα σύστημα και αναγνώρισης προσώπου, το οποίο ίσως είναι το πιο εύκολο στην αξιοποίησή του, παρουσιάζει ωστόσο μειονεκτήματα, διότι μπορεί να προκύψουν διαφορές ως προς το ε, πρόσωπο που επαληθεύεται από το μηχάνημα σε σχέση με μια φωτογραφία που έχει καταγραφεί στο σύστημα. Φερρυπίν άφησε μουστάκι ή άφησε μουσια και παρουσιάζει διαφορά. Άρα στα συστήματα διαχείρισης συνόρων δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε ένα σύστημα αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει αποδεδειγμένα το μικρότερο ποσοστό λάθους και είναι αυτό των δακτυλικών αποτυπωμάτων, συμπληρωματικά. Με ένα δεύτερο λοιπόν βιομετρικό σύστημα πέραν της αναγνώρισης προσώπου. Εμείς έχουμε εισαγάγει στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, τέτοια συστήματα και σκοπεύουμε στο μέλλον να εισαγάγουμε πέραν της αναγνώρισης τακτιλικών αποτυπωμάτων και αυτό της αναγνώρισης προσώπου. Αντίστοιχα προσβλέπουμε σε διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες που μπορούν να αξιοποιήσουν έτσι αυτά τα συστήματα επικοδομητικά. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετοιμάσει ένα σύνολο προτάσεων για τα εφη σύνορα εισόδους εξόδων, εισόδους εξόδους στο σύστημα Schengen. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να διευκολύνει ιδιαίτερα ε, τη διακίνηση Τούρκων επικών και δι επιχειρηματιών ή ανθρώπων του πνεύματος, ε, καθηγητών και ούτω καθεξής, που τακτικά θέλουν να ταξιδεύουν στις χώρες Σέγγεν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων πιστεύω ότι μπορεί να μας επιτρέψει χάρη και στο σύστημα ΙΠΑ, στο προενταξιακό δηλαδή μέσον, που άλλωστε έχουμε αξιοποιήσει στα προηγούμενα χρόνια σε συνεργασία με χώρες γειτονικέ και όμορες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Έχουμε λοιπόν αξιοποιήσει το ε, προταξιακό μέσον είπα για να αναπτύξουμε καλύτερη διαχείριση των κοινών μας συνόρων και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον αυτή την προσπάθεια. Το Frontex ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των εξωτερικών συνορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνεχίζει την ε, καταγραφή των νομοθετημάτων και σε ό,τι αφορά την Τουρκία έχουμε για το 2011 και το 2012 στο πλαίσιο του προενταξιακού μέσου είπα, συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας όπως το Βαν, το Χάκιαρι και άλλες όπου στόχος μας είναι και η χρηματοδότηση του ΕΠΑ προβλέπει την ε, αφαίρεση ναρκών και τον καθαρισμό των παραμεθοριών περιοχών. Επίσης, με συμμετοχή και συνεργασία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ε, και αντίστοιχων φορέων έχουμε προχωρήσει σε σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, ναρκωτικών, της λαθρέας διακίνησης ανθρώπων. Έχουμε ετοιμάσει τη σχετική νομοθεσία και έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία σε διάφορες πλατφόρμες όπου η Τουρκία πιστεύω μπορεί να αποδείξει πως είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα συστήματα ολοκληρωμένων σύνορων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής. Κυρία Πρόεδρε, ε, με τη σειρά μου να καλωσορίσω και εγώ τα μέλη των εθνικών ε, αντιπροσωπιών, των κρατών μελών που βρίσκονται μαζί μας. Ε, να ευχαριστήσω την κυρία Φαγιόν και τον κύριο Ντεμέρα για τις εξαιρετικές εισηγήσεις τους που φαίνεται ότι με πολύ ωραίες συναντήσεις έχουν κάνει πολύ οργανωμένη και εξαιρετική δουλειά. Την κυρία Υπουργό, τον κύριο Επίτροπο που δεν μπόρεσε να παραμείνει περισσότερο Θέλω να προσθέσω ε, δύο σκέψεις με συντομία πάνω σε όσα υπόθηκαν και παίρνοντας αφορμή και από την τοποθέτηση του κυρίου Κοέλιου που είχε ασχοληθεί εξαιρετικά πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε. Πράγματι, αυτό που μας απασχολεί είναι η στόχευση μιας νέας νομοθετικής πρότασης. Γιατί θέλουμε είναι μόνο διότι πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο τα εξωτερικά μας σύνορα και αν συμβαίνει αυτό τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει και το βιώνουμε όλοι είναι ότι λόγω των γενικότερων ανακατατάξεων σε χώρες ε, όμορες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες όπου ε, διαπιστώνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα υπάρχει μια ανεξέλεγκτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά έχει διαφοροποιηθεί το πολύ σημαντικό θέμα της τρομοκρατίας με την έννοια της αλλαγής των κινήτων και των τρόπων δράσης των οργανωμένων αυτών ομάδων και βεβαίως το διασυνοριακό έγκλημα το οποίο έχει λάβει τη μορφή εγκληματικών οργανώσεων διεθνικού χαρακτήρα και αυτό πάλι ε, με διάφορες μορφές εκτέλεσης και εκδήλωσης δεν ελέγχεται. Αυτή είναι η στόχη υπάρχουν δύο παράλληλοι διάλογοι από ό,τι κατάλαβα και από τις δύο εισηγήσεις της κυρίας Φαγιών και του κυρίου Ντεμέρα. Ο διάλογος ο ένας αφορά στην κοστολόγηση ενός τέτοιου οργανωμένου συστήματος ελέγχου των εξωτερικών συνόρων προωθημένου. Αυτός ο διάλογος βέβαια φαντάζομαι ότι θα διεξαχθεί και με τη συμμετοχή πολλών τεχνοκρατών οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ο δεύτερος διάλογος αφορά στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ε, το, το θέτω, διότι όπως και στη, στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται, θα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να λάβουμε όλες τις εθνικές νομοθεσίες που υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από κράτη σε κράτη. Οι αποκλίσεις βέβαια δεν είναι τέτοιες ώστε να μας διαφοροποιούν για την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των ελευθεριών. Φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Για την ανάγκη κατοχύρωσης της συλλογής των δεδομένων στα πλαίσια της οργάνωσης του συστήματος. Εκεί θα πρέπει με τον προωθητικό διάλογο να αποφασίσουμε ποια στοιχεία θα συλλέγονται, από ποιους θα συλλέγονται, ποιοι θα έχουν πρόσβαση και για ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συντηρούνται ούτω ώστε να καταχειρώνονται παράλληλα οι ελευθερίε, οι προσωπικέ ελευθερίε. Σε αυτό, νομίζω σε αυτό το δεύτερο τμήμα του διαλόγου θα είναι πολύ χρήσιμα αυτά που ανέφερε η κυρία Φαγιόν για τα 12 κράτη-μέλη που έχουν πιλωτικά συστήματα, τα συμπεράσματα από τη χρήση αυτών των πιλωτικών συστημάτων φαντάζομαι ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στο διάλογο και στην σύγκληση των διαφορετικών απόψεων που πάντως δεν θα είναι θεσμικές, θα είναι λειτουργικές περισσότερο από κράτος σε κράτος. Αυτές τις ε, επισημάνσεις ήθελα να κάνω και βέβαια ε, να πούμε ότι σε αυτό το διάλογο που ξεκινάει δεν είναι μόνο δεν μας αφορά μόνο όπως προείπα το γεγονός ότι διευρύνθηκαν τα σύνορά μας γιατί αυτό στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι ότι θέλουμε μια Ευρώπη με ανοιχτά σύνορα ελεγχόμενα μεν αλλά όχι μια Ευρώπη φρούριο στην οποία κανείς δεν θα έχει πρόσβαση το αντίθετο και ξέχασα μόνο να πω ότι στις παραμέτρους που έχουν συμβάλει τα τελευταία χρόνια για να έχουμε την αναγκαιότητα να μελετήσουμε ένα νέο σύστημα ε, διαφύλαξης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων είναι η παράτυπη μετανάστευση ο έλεγχος της οποίας είναι η πραγματική οδός για την κατοχήρωση της νόμιμης μετανάστευσης, εκεί όπου συμβάλλει και στην Ευρώπη για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας και ε, αναχώρα στην αναλογική κατανομή τέτοιων ανθρώπων, ιδιαίτερα με ειδικέ ε, τεχνογνωσίες, που είναι χρήσιμες για την εξέλιξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, δεν έχω άλλο κίτρινο έντυπο, αλλά ναι, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κόμες, Ευρωβουλευτής από τους Σοσιαλιστές, την ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή και τους εισηγητές μας βέβαια κάτι. Κάτι που θα έλεγα ότι έρχεται πριν από τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του συστήματος το θέμα της αναλογικότητας, αναγκαιότητας κτλ. Είναι σαν να επικεντρωνόμαστε πολύ στο θέμα της ροής των μεταναστών, αλλά τι γίνεται με τους πλούσιους μετανάστες που τελικά είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία κτλ. με το πακέτο αυτό εξετάζουμε και καταστάσεις που γνωρίζουμε ότι οδηγούν στην είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατόμων που ενδυνάμει είναι εγκληματίες. Το θέμα των Golden Visit είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή δεν ήθελε να ασχοληθούμε με αυτό γιατί λέει ότι είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Μα όταν μιλάμε για ευφύ σύνορα, Όσοι έχουν άδειε παραμονής, προφανώς και θα μετακινούνται συχνά, αλλά τι επίπτωση θα έχει αυτό. Τώρα, για αυτές τις χρυσές θεωρήσεις, είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους οι χώρες. Αλλά μήπως με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε εγκληματικότητα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι κάτι που έχει να κάνει με την έρευνα που έγινε από τις πτήσεις της CIA. Όταν έχουμε να κάνουμε με ιδιωτικές πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι έλεγχοι είναι πολύ περιορισμένοι σε αυτούς που φτάνουν με τέτοιες ιδιωτικές πτήσεις, ανύπαρκτη θα έλεγα, ενώ οι επιπτώσεις για την προστασία των συνόρων μας είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε μια χώρα μέλος χωρίς έλεγχο. Πάντα πρόκειται για τους πλούσιους βέβαια, έτσι, που έρχονται με τα ιδιωτικά τους αεροσκάφη. Έχουμε σκεφτεί καθόλου πώς συνδυάζεται αυτό με τα ευφύ σύνορα. Αυτές λοιπόν είναι δύο ερωτήσεις που νομίζω ότι θα έπρεπε να εξεταστούν πριν περάσουμε στο θέμα των τεχνικών προδιαγραφών και του κόστους του πακέτου αυτού ευφύ σύνορα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μελό τελευταίος από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μέλο. Θέλω να σας πω ότι είμαι απολύτως υπέρ του συστήματος αυτού έφη σύνορα. Η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η τρομοκρατία. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα που αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά αυτό το σύστημα εισόδων-εξόδων και το θέλουμε. Γιατί εμείς βλέπετε έχουμε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε Συνεπώς να αντικαταστήσουμε ένα παλιό απαρχιωμένο σύστημα και να προσαρμοστούμε με ένα νέο σύστημα που με τη σειρά του να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ε, σημερινές ε, ανάγκες. Με ρομαντισμό δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές λέμε ότι τίθεται ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εννοείται ότι πρέπει να το προσέξουμε αυτό τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η προστασία της ζωής, το δικαίωμα στη ζωή. Δεν είναι λιγότερο σημαντικό δικαίωμα, δεν χρειάζεται κανείς να είναι νομικός για να το αντιληφθεί αυτό. Στις σχολές νομικής πάντως πρέπει να σας πω ότι εμείς το μαθαίνουμε αυτό το θέμα της σύγκρουσης δικαιωμάτων. Υπάρχει μια ιεράρχηση δικαιωμάτων, δηλαδή κάποια δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από άλλα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2013, πάνω από 16 εκατομμύρια θεωρήσεις δόθηκαν για μικρής διάρκειας παραμονή και πάρα πολλές άλλες αιτήσει απορρίφθηκαν. Σε μερικές περιπτώσεις όμως διαπιστώσαμε ότι τα άτομα αυτά είχαν καταφύγει στην απάτη και ότι τελικά είχαν πλαστογραφήσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Όσον αφορά τώρα τους ελέγχους στα αεροδρόμια, από τα 400 εκατομμύρια και θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός στο μέλλον. 0,9% των ατόμων που μπαίνουν τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθούν να βρουν δουλειά ή έρχονται για τουρισμό ή επισκέφτονται συγγενείς τους. Υπάρχει όμως και το υπόλοιπο που είναι μικρό μεν ποσοστό, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν απειλή και μπορούν να προκαλέσουν πραγματικές τραγωδίες στις χώρες μας. Οπότε, μερικές σαφείς ιδέες ή ερωτήσεις άμα θέλετε. Στον κώδικα του Σέγγεν δεν προβλέπονται προδιαγραφές για τη διέλευση. Μόνον η σφραγίδα ε, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε η σφραγίδα στο διαβατήριο πότε μπήκανε και πότε βγήκανε. Σωστά. Δεύτερον, τα σύνορα στα σύνορα υπάρχει βάση δεδομένων για την είσοδο, όχι όμως και για την έξοδο. Οπότε δεν γνωρίζουμε πότε βγήκανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα αυτά. Και τρίτον, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και εθνικά δεδομένα για να εντοπίσουμε άτομα τα οποία έχουν παραμείνει περισσότερο στις χώρες μας από ό,τι επιτρέπεται βάσει της άδεια που έχουν. μπορούμε να ελέγξουμε, να συγκρίνουμε και να γνωρίζουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα εθνικά δεδομένα και εντοπίσουμε τέτοιες αναντιστοιχίες, τι γίνεται στη συνέχεια. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ερωτήσεις που με προβληματίζουν και γι' αυτό και τις εκφράζω, γιατί κατά τα άλλα σαφώς και είμαι υπέρ αυτού του πακέτου μέτρων για πιο ευφυή σύνορα δεδομένη στη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Μάκερ, ευχαριστώ. Όσον αφορά τα ευφύ σύνορα, για να μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε σύνορα. Η Ευρώπη στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, διότι είναι διάτρητα τα σύνορα. Το σύστημα αυτό θέλουμε να το βελτιώσουμε, να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση και να προστατευτούμε καλύτερα. Ερώτηση μου λοιπόν στους ηγητές και στην Επιτροπή είναι εξής. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι παράνομοι μετανάστες και οι εγκληματίες οι οποίοι παίρνουν χιλιάδες ε, χιλιόμετρα για να φτάσουν στις χώρες μας. Πιστεύετε ότι μέσω ενός τέτοιου ηλεκτρονικού συστήματος θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να μην μπουν τελικά στις χώρες μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε λίγα λεφτά στη διάθεσή μας τώρα για απαντήσεις. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Φαγιόν και στον κύριο Δία Ντεμέρα, στους δύο συγκητές μας δηλαδή, για να απαντήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές σας ερωτήσεις και ομιλίες. Ακούγοντάς σας όλους, συμπέρανα κάποια περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω λοιπόν μαζί σας πρώτον το εξής. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό κίνδυνο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Όλοι πιστεύουμε ότι απαιτούνται ε, να υπάρχουν ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα συστήματα σήμερα με τον σωστό τρόπο και το EES και το CES χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο πριν αρχίσουμε να συζητάμε την εφαρμογή του νέου συστήματος στα σύνορα. Πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο πραγματικός στόχος των συστημάτων αυτών για τα ευφυή e σύνορα. Θυμάστε ότι στην αρχική πρόταση μιλούσαμε για κάποια διευκόλυνση αλλά τώρα συζητάμε και ξεκάθαρα και για το θέμα της πρόσβασης των αστυνομικών αρχών, των αρχών επιβολής ε, ε, της τάξης και τα λοιπά, ε, είναι ένα επιπλέον θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε κάνει κάποια πρώτα βήματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία και τα κράτη-μέλη. Ακούσαμε όμως για μια ακόμη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες αυτές τις ανησυχίες που θα οδηγήσουν σε μια νέα πρόταση στις αρχές του 2016. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει μια αναθεωρημένη πρόταση. Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόταση αυτή όταν αποσυρθεί στο τέλος του χρόνου η πρόταση που ισχύει σήμερα. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα, θα παραμείνει σε ισχύ. Έχουμε μια πιλωτική φάση σε ορισμένες χώρες, σε 17 μεθοριακά σημεία. Ελέγχουμε αν θα πρέπει να έχουμε 4 ε, ε, δακτυλικά αποτυπώματα, 10 δακτυλικά αποτυπώματα και άλλες τεχνικές λύσεις. Το Νοέμβριο θα έχουμε στη διάθεσή μας την τελική έκθεση. Έχουμε επενδύσει αρκετά χρήματα και γι' αυτό θα περιμένουμε τότε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ανησυχίες μου όμως είναι υψηλέ. Θα ήθελα να γίνουν σοβαρές συζητήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Γιατί πάρα πολλές ερωτήσεις και μάλιστα καλές ερωτήσεις ε, δεν μας δίνουν στοιχεία για την ε, ε, τη σχέση κόστους-οφέλους ε, και επίσης ε, για το τι θέλουμε. Θέλουμε να διευκολύνουμε το πέρασμα των συνόρων ή θέλουμε να καταστήσουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ε, και επισκέπτες υπόπτους. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία λαμβάνουμε στην Ευρώπη και δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό χωρίς να αποκαταστήσουμε την ισορροπία με την βασική έννοια που είναι η ελευθερία της κίνησης. Και ε, πόσα χρήματα θέλουμε να ξοδέψουμε στα νέα συστήματα αν δεν χρησιμοποιούμε πλήρως τα παλιά συστήματα. Αυτά λοιπόν συγκράτησα από τους προηγούμενες ομιλίες και αυτά είναι τα θέματα που θα ήθελα να θέσω κι εγώ. Ευχαριστώ Τάνιο. Ο κύριος Διεστεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω, όχι απλά, αλλά θα προσπαθήσω να συνθέσω τις απαντήσεις μου για να καλύψω όλες τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. 13 άνθρωποι πήραν το λόγο, 13 βουλευτές. Οι περισσότεροι ήταν εθνικοί βουλευτές και οι υπόλοιποι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις Πορτογάλοι μάλιστα από τους ευρωβουλευτές. Δείχνεται, δι, φαίνεται έτσι πόσο ζωντανή είναι αυτή η χώρα και πόσο διαφορετικές απόψεις επικρατούν εκεί. Όλες αξιοσέβαστες. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνατε. Πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια παλιά νομοθετική πρόταση για την οποία ακούστηκαν διάφορες επικρίσεις γιατί δεν ήταν σαφής ο στόχος, δεν υπήρχε σαφής ορισμός του στόχου και γι' αυτό το κόστος ήταν πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αυτά αρχικά. Τώρα, μας ήρθε η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα θέλει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως του αντιστοιχεί μια που είναι συνομοθέτης, προκειμένου να επηρεάσει αυτό το νομοθετικό πακέτο που αποτελείται από τρεις εκθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα προχωρήσει σε νέα νομοθετική πρόταση αφού έχει εξολογήσει την τεχνική έκθεση που την έχουμε, 600 σελίδες στα αγγλικά, και από την άλλη μεριά τα συμπεράσματα της δοκιμαστικής περίοδου. Τι λέει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι λέμε η Τάνια και εγώ που είμαστε οι κύριοι συγητές. Λέμε όχι. Πριν το Κοινοβούλιο προχωρήσει στην ε, δικιά του νομοθετική πρόταση, του 2016 δηλαδή, ε, το είπαμε στον κύριο πρέπει πρώτα να ακούσουμε τους ευρωβουλευτές μας και να ακούσουμε και τους εθνικούς βουλευτές. Αυτή είναι η αρχή λοιπόν σήμερα, γιατί θα υπάρξει και συνέχεια, σαν τη σημερινή συνεδρίαση δηλαδή, για να ακούμε και τη φωνή των εθνικών βουλευτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Τάνια, ότι στις αρμόδιες εθνικές κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία κάνει πρόταση χωρίς να λάβει υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, για την νομοθετική πρόταση έτσι αλλιώς πρέπει να περάσει από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πρόκειται για συναπόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τώρα, τι ισχύει. Προσοχή, μην μπερδεύουμε τους στόχους. Και αυτό το λέω κυρίως στους συναδέλφους μου ευρωβουλευτές. Μην μπερδεύετε τους στόχους. Να εντοπίσετε καλά ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της πρόταση αυτής και ποιοι είναι οι δευτερεύοντε στόχοι. Δεν θέλω να σας κουράσω και να πω όσα είναι ήδη γνωστά. Μην μπερδεύετε τους στόχους όμω. Και εδώ επαναλαμβάνω ότι πέρα από αυτά που λέω εγώ όσον αφορά την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου, αυτό είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Αυτό που λέω εγώ δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση που πρόκειται να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ μπορεί να έχω τη δικιά μου τη θέση, αλλά δεν σημαίνει ότι θα περάσει αυτή. Ελπίζω να είναι και η άποψη της πολιτικής μου ομάδας. Αλλά όχι να ρίχνουμε το ανάθεμα τώρα για το κόπο. Το είπε και ο κύριος Αφραμόπουλος πριν, πολύ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει απόφαση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι λέει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωραία, ρίχνει την πρότασή της. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όμως θα αποφασίσουμε. Και η συνέχεια, αυτά τα οποία απασχολούν εσάς και αυτά που απασχολούν εμάς, τους δύο εισηγητές. Απλοποίηση πρώτον, κόστος δεύτερον. Απλοποίηση όσον αφορά την προστασία δεδομένων, να έχουμε ένα σύστημα διέλευσης ε, συνόρων που να συνοδεύεται από σύστημα προστασίας των δεδομένων. Τρίτον, το θέμα της διαλειτουργικότητας, δηλαδή να εποφεληθούμε από αυτά που έχουν ήδη τα κράτη-μέλη, να τα εμπλουτίσουμε με την τεχνική έκθεση και να λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα της δοκιμαστικής περίοδου. Μιλάμε για βελτίωση των ελέγχων στο, στα σύνορα. Αυτά που ρώτησε ο Νούνο το είχε απαντήσει ο Επίτροπος Αβραμόπουλος. Είναι τα βασικά. Το σύστημα, το σημερινό, οι σφραγίδες δεν φτάνουν. Ξέρουμε πότε μπαίνει κάποιος στα σύνορά μας, δεν ξέρουμε όμως πότε βγαίνει. Αν μείνει 60, 90 ή τις ξεπεράσει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εφόσον δεν ξέρουμε και την είσοδο και την έξοδο του ατόμου. Οπότε, ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να ακούσω και την Τουρκία. Τι είπε. Γιατί είναι μια μεγάλη χώρα η Τουρκία. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, τεράστια, που έχει μεγάλη ισχύ όσον αφορά την ε, ασφάλεια της Ευρώπης. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα δώσουμε πρόσβαση στο σύστημα στις αρχές ασφάλειας. Είχατε την ευκαιρία να πείτε αυτά που είπατε, εντάξει, μου πετάξατε το γάντι και σας το επιστρέφω. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα τόσο σημαντική και τόσο ισχυρή όπως είναι η Τουρκία, να μην επιτρέπει την ε, μετακίνηση ξένων μαχητών για να πάνε στο κομπάνι. Πρέπει να βοηθάτε με πληροφορίες τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Σήμερα και αύριο η Τάνια και εγώ θα συγκεντρώσουμε τα στοιχεία από τις παρεμβάσεις σας και θα συνοψίσουμε στο τέλος. Με προσωρινά συμπεράσματα. Προς το παρόν είμαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ Κυρία Σιλίνια, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε, πιστεύω, με τους αδέλφους ότι όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους δευτερεύοντες στόχους υπάρχει όμως σαφής συμφωνία ότι θα, πει, θα υπάρχουν πάντα πρώτα πρωτεύουσα σημασία και δευτερεύοντα ζητήματα. Από πολλού όμω από του ομιλητέ ε, ακούω ότι δεν λειτουργεί αποτελεσματικά το υφιστάμενο σύστημα και δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τα εντυνόμενα προβλήματα της επικαιρότητα όπως την εντυνόμενη μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση, τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Ανέφερε και η κυρία Ρόζενπερ και επί ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα όπως το οργανωμένο έγκλημα και άλλα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά. Αυτό νομίζω μπορούμε να το δούμε με την νέα πρόταση που περιμένουμε να κατευθεί σε σχέση δε και με την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Με χαρά σημειώνω ότι θα απαιτηθεί αξιολόγηση για την υποβολή προτάσεως των ευφυών συνόρων ή πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου παράλληλα με το, η συζήτηση για το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση θέλουμε βεβαίως να γίνεται αλλαγή απόψεων και θα συνεργαστούμε ενεργά με τους συνεισηγητές. Συμφωνούμε πως οι νέες τεχνολογίες είναι ένας τρόπος αξιοποίησης αποτελεσματικότερα των συστημάτων, των συνόρων και εντοπισμού των, ή αναγνώριση καλύτερα των προσώπων που διέρχονται και περιορισμού βέβαια του διασυνοριακού εγκλήματος. Προς το παρόν αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ξέρω ότι θα είναι εύκολο να αντικαταστήσετε τον κύριο Βρωμόπουλο σήμερα, αλλά μια και έχουν διατυπωθεί πολλές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Θα προσποιηθώ ότι είμαι ο κύριο Αβραμόπουλος, λέει η κυρία Φάικ. Πάνω απ' όλα για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Με στοιχεία κυρίω Έχουμε 1800 φυλάκια συνοριακά. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη γιατί αύριο θα ακούσουμε συγκεκριμένα για τη ζωή των ανθρώπων αυτών που δουλεύουν οι συνοριοφύλακες θα μας δώσουν μια εικόνα του τι σημαίνει η διαχείριση αυτών των ε, φυλακίων και επίσης εν γέννη για τα συστήματα εισόδου-εξόδου έχουν αξία γιατί μπορούμε να καταγράφουμε αν κάποιος μπήκε από ένα μέρος και βγήκε από ένα άλλος. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία με 1800 συνοριοφυλάκια. Έχουμε 600 δε εκατομμύρια διαλέψεων, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια ήταν διαλέψεις από υπηκόους τρίτων κρατών, όπως είπε και ο Επίτροπος. Με επιτυχία σημειώνουμε, χωρίς ε, παρανομία, 100.000 ήταν αυτοί το, στους οποίους απορρίφθηκε η είσοδος, η η είσοδος στα σύνορα και είχαμε παράνομες εισόδους περί τις 280.000. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν τα σύνορά μας καλά, λειτουργούν αρκετά καλά με όσες ανάγκες και αν υπάρχουν για βελτίωση. Τα συστήματα τα οποία ε, συζητούμε αφορούν τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος Schengen. ο τρόπος με τον οποίο όμως διαχειριζόμαστε τα σύνορά μας, ποιος δηλαδή, σημαίνει το ποιος θα είναι δεκτός, ποιος μπορεί να μπει στο σύστημα Schengen, ποιος θα λαμβάνει την άδεια εισόδου. Επίσης θέλω να σημειώσω γιατί ο χρονισμό των νέων προτάσεων. Είπε ο Επίτροπος ότι στοχεύουμε στις αρχές του 2016 να κατεθεί νέα πρόταση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το χρόνο να αξιοποιήσουμε και τα αποτελέσματα των πιλωτικών, των δοκιμαστικών αυτών εφαρμογών που θα συζητηθούν και αύριο περισσότερο το γιατί δεν αποσύρεται η φυστάμενη πρόταση οφείλεται στο ότι ε, δίνει αξία στην ε, λύση ο Επίτροπος. Ξέρουμε ότι συζητούμε πάνω σε προτάσεις που θα αλλάξουν, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά προτιμούμε να διατηρήσουμε την παλαιά πρόταση, γιατί αν πρόκειται η είσοδος-έξοδος και οι καταχωρημένοι ε, ταξιδιώτες να συγχωνευτούν σαν έννοια, θα είναι καλό να έχουμε στη, σαν βάση ένα κείμενο, έστω και αν αυτό δεν ισχύει. Επίσης για την νομοθετική πρόταση θα γίνει αξιολόγηση συνοποιών όχι μόνο για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θα αφορά μόνο αυτό η αξιολόγηση συνοποιών, Αλλά θα, θα αντιμετωπιστεί και αυτό. Θα γίνει αξιολόγηση συνοποιών, λοιπόν, όπως έγινε και για την υφιστάμενη πρόταση. Τα θετικά και τα αρνητικά τα έχουμε καταγράψει. Τα σημαντικά, πολύ σημαντικά πλονεκτήματα για την πρόσβαση των αρχών επιβολή του νόμου στο στόχο, το σημαντικό στόχο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά βέβαια και στα αρνητικά της προσβολές ή τα αρνητικά στοιχεία τα σχετικά με την προσοχή των προσωπικών δεδομένων. Το 2013 ελήφθη η απόφαση ότι δεν ήταν κατάλληλη στιγμή για την επιβολή της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου όπως άλλωστε και για τη θεώρηση των διαβατηρίων. Σημειώνουμε τι τοποθετήσει των Διεθνικών Κοινοβουλίων, τις συστήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ληφθούν υπόψη και θα τροφοδοτήσουν την αξιολόγηση συνεπειών, χωρίς να μπορώ βεβαίω να προδικάσω το τι θα πει η τωρινή Επιτροπή ε, για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Θέλω να σημειώσω ότι υπήρχε η αξιολόγηση θετική αλλά και με κάποια αρνητικά στοιχεία από την προηγούμενη Επιτροπή της Πρόσβασης των Αρχών Επιβολής του Νόμου. Ε, θέλουμε όσο το δυνατόν να έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα στο νέο σύστημα. Το σημειώνουμε, επί παραδείγματι, στην ε, διατή έκθεση διαχείριση Schengen. Επίσης, κάνουμε αξιολόγηση του συστήματος πληροφοριών Schengen αναμένεται του χρόνου αλλά και ενδιαμέσως αν υπάρξουν κάποια στοιχεία θα σας τα διαθέσουμε γιατί είναι απαραίτητο να τα έχουμε στη θέση μας το ταχύτερο δυνατό. Για το θέμα κόστους και προϋπολογισμού δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ξέρετε ότι το Ταμείο για την Ασφάλεια έχει προβλέψει 791 εκατομμύρια κατά μέγιστον ευρώ. Με στοιχεία δεν περσινά βλέπουμε ότι το κόστος ενός ενιαίου συστήματος περιορίσουμε σημαντικά τη δαπάνη από χωριστά εθνικά συστήματα ή άλλες τεχνικές επιλογές. Πάντως θα χρειαστεί να προβλεφθεί ο σχετικός προπολογισμό για να καλυφθεί και το κεντρικό κόστος ανάπτυξης και διαχείρισης σε λειτουργία του συστήματος, του κεντρικού συστήματος, αλλά και εκείνο το κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία των εθνικών συστημάτων. Πολλά δίνεται διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Το κύριο και Πρώτο είναι ότι δεν ξεκινάμε να, να χρηματοδοτούμε σύστημα αν δεν ξέρουμε τι θέλει να ε, εξυπηρετήσει. Δεν αρχίσουμε να το φτιάχνουμε αν δεν ξέρουμε τι στόχο εξυπηρετεί. Το είπε και ο κύριος Κουέλιο. Και επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι αντιληφθήκαμε τι είδου συνέπειε μπορεί να ή να αντιλαμβανόμαστε τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει κάθε νέο σύστημα στα εθνικά συστήματα. Αυτό δεν ήταν και για πολιτικούς λόγους δυνατόν με την εισαγωγή του ΣΥΣ. Ε, και ξέρουμε ότι κόστησε πολύ ακριβά στα κράτη. Ε, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μια σωστή αντίληψη των συνεπειών τόσο για το κεντρικό όσο και για τα εθνικά συστήματα. Αυτές πιστεύω ήταν οι κύριες παρατηρήσεις. Και υπογραμμίζω ότι οι πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν πρωταρχική σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα, πάντα αφορούν τους υπηκόους τρίτους κρατών με τα ίδια, με το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως και για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουν σημαντική επίπτωση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα μέτρα γιατί θα προσδιορίζουν διαφορετικό χρόνο διέλευση στο χώρο Σέγγεν και βεβαίως θέλουμε οι υπήκοοι τρίτων κρατών να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα υπάγονται στη διαχείριση του συστήματος υπηκοή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι ηλεκτρονικές θύρες πιστεύουμε ότι θα διευκολύνουν τους πάντες. Και κυρία Γκόμες, λυπούμε, αλλά νομίζω ότι ξέχασα τη δική σας ερώτηση. Διατυπώστε το ίδιο ερώτημα με την προηγούμενη φορά. Τι γίνεται με την χρυσή λεγόμενη θεώρηση. Για να απαντήσω συνοπτικά, πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δεν έχουμε αρμοδιότητα ως Επιτροπή. Αλλά θα ε, ζητήσω, θα υπερθυμίσω στον Επίτροπο να σας αποστείλει χωριστή απάντηση. Είναι ένα θέμα χωριστό από αυτό των ευφύων συνορών, αλλά αντιλαμβάνομαι την πολιτική σας επισήμανση. Για μας και κατά τη δική μας θεώρηση, το σύστημα ισχύει για τους πάντες, πλούσιους ή φτωχούς. Τα πάντα τα εξαρτώνται από το μέσον με το οποίο καταφθάνουν στα σύνορα. Αλλά ίσως αύριο να συζητηθεί και από τους συναδέλφους που θα μιλούν για, τα, για τις διελεύσεις το ζήτημα των ιδιωτικών αεροσκαφών ή ιδιωτικών θαλαμιγών. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Προεδρία, εισηγητές, συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλους όσοι έλεγαν το λόγο σήμερα. Θα διακόψουμε για λίγο, θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά μόνο καλό τους συναδέλφους που πρόκειται να λάβουν το λόγο για το επόμενο κομμάτι της συζητήσεως να έρθουν στο Προεδρείο. Good afternoon. Um, if we can start uh, our session, uh, I say good afternoon and hello. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους. Θα ομιλήσω την ρωμανική. Βάλτε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα ήθελα να πω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει ανάγκη από ένα βιώσιμο και σύγχρονο σύστημα ελέγχου των συνόρων. Και νομίζω ότι το Σέγγεν μπορεί να αποτελέσει μία λύση. Το Σέγγεν δεν είναι το πρόβλημα. Βασιζόμενοι λοιπόν στα μέσα τα οποία μας δίδει το κοινοτικό κεκτημένο, και αποκαλούμεθα να ενισχύσουμε άλλωστε, θεωρώ ότι το σύστημα Schengen είναι η καλύτερη λύση για να ασκήσουμε τις θεμελιώδεις μας, τα θεμελιώδη μας δικαιώματα. Είναι καθήκον μας ε, να μην ε, υπακούσουμε στις σιρήνες του λαϊκισμού Ξέρουμε τι σημαίνει το Σέγγεν για την ασφάλεια του Ευρωπαίου πολίτη και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η Ρωμανία δεν είναι μέλος του χώρου Σέγγεν αλλά έχει αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του συστήματος. Από τον Νοέμβριο μάλιστα του 2010 το κάνουμε αυτό. Είμαστε μέλη επίσης και στο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αναφέρθηκε λίγο προηγουμένως στην ουσία εμείς δρούμε σαν de facto μέλος του χώρου Σέγγεν και συνεισφέρουμε στην βελτίωση της ασφάλειας των κρατών μελών. Με βάση λοιπόν τις συγκεκριμένες αυτές παρατηρήσεις θα κατανοήσετε αυτή την αίσθηση αδικίας την οποία έχουμε εμείς και τη δυσφορία που νιώθουμε όταν φτάνουμε στον χώρο Σέγγεν και κάθε φορά Πρέπει να υποβληθούμε σε πολιτικού τύπου κριτήρια ελέγχου και όχι σε κριτήρια τεχνικά όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδριάσεως οι συζητήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ελπίζω λοιπόν ότι και αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρόζενμπουργκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας ενημερώσει για την τεχνική μελέτη που έγινε πέρυσι. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ρόζενμπεργκ, να προσκαλέσω όλα τα μέλη που θέλουν να πάρουν μέρος στην συζήτηση να δηλώσουν το όνομά τους το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα στοιχεία τους και να επιτρέψουμε μια δίκαιη θα έλεγα συζήτηση στη συνέχεια. Κύριε Ρόζεμπουργκ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπλήρωσε την τεχνική της μελέτη για τα ευφύ σύνορα τον Οκτώβριο του 2014. Ήδη παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ της 16ης Οκτωβρίου του 2014. Το κεφάλαιο για το κόστος παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο και έγιναν και άλλες ε, τεχνικές συναντήσεις από τότε. Η μελέτη είναι διαθέσιμη online, είναι άνω των 600 σελίδων. Αυτά τα οποία θα σας πω τώρα δεν είναι νέα για πολλούς από σας, όμως ε, θα σας θυμίσω κάποια στοιχεία βασικά ε, από τα ευρήματα στα οποία καταλήξαμε ε, και βέβαια θα τα πω συνοπτικά γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Είναι το πρώτο βήμα της λεγόμενης αποδεικτικής επίδειξης της μεθόδου την οποία συμφωνήσαμε με τους συνεισηγητές τον Φεβρουάριο του 2014. Το δεύτερο τμήμα είναι η φάση τεστ ελέγχου στην οποία θα έρθω αργότερα. Έγιναν οι αρχικές προτάσεις το 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έθεσαν θέματα τεχνικά, λειτουργικά και κόστους. Ε, στόχος της μελέτης ήταν να δώσουμε απαντήσεις στις απορίες αυτές όχι στα θέματα τα πολιτικά βέβαια, αλλά στα θέματα τα τεχνικά, τα πρακτικά. Η μελέτη λοιπόν κάνει μία ανάλυση με απαντήσεις ε, σε τέσσερις ομάδες θεμάτων. Καταρχάς στην αρχιτεκτονική του συστήματος, στα βιομετρικά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, στα θέματα της συλλογή δεδομένων, και στα θέματα των μεθοριακών ελέγχων και τις διαδικασίες. Το πέμπτο θέμα, το κόστος, είναι κάτι που αφορά όλα τα προηγούμενα. Για την πρώτη διάσταση, για την αρχιτεκτονική του συστήματος. Ήδη οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 παρουσίασαν δύο διαφορετικά συστήματα, το EES και το RTP. Η μελέτη αποδεικνύει ότι είναι προτιμότερο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα το οποίο να περιλαμβάνει τις λειτουργίες του EES και του RTP. Αυτό θα μειώσει το κόστος ανάπτυξης, θα αποτρέψει τις επικαλύψεις και θα μειώσει τις επιπτώσεις στα εθνικά συστήματα. Ένα ενιαίο σύστημα θα είναι και ευθυνότερο από ό,τι δύο ξεχωριστά και το είχαμε πει και το 2013. Η διαφορά είναι σημαντική, 49 εκατομμύρια στα 4 χρόνια. Ένα άλλο θέμα το οποίο η μελέτη εξετάζει είναι η σύνδεση ανάμεσα σε αυτό το νέο ενιαίο σύστημα από τη μία και στο σύστημα ενημέρωσης ε, θεωρήσεων ε, του Σέγγεν από την άλλη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε εδώ ότι όπως προβλέπαμε και στις προτάσεις του 13 το ESRTP και το σύστημα ενημέρωσης των θεωρήσεων θα χρησιμοποιούν ένα κοινό βιομετρικό σύστημα αντιστήχησης, το BMS. Το ESRTP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά πληροφορίες από το VIS, το σύστημα δηλαδή ε, ε θεωρήσεων, και αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα μεταξύ τους θα είναι διαλειτουργικά, θα μπορεί να συνομιλεί το ένα με το άλλο. Σχετικά με την παρούσα αρχιτεκτονική των συστημάτων έχουν αναλυθεί τρεις βασικές επιλογές. Καταρχάς ένα ESRTP ανεξάρτητο από το σύστημα θεωρήσεων. Δεύτερον ένα ESRTP ενσωματωμένο στο VIS, το σύστημα ενημέρωσης των θεωρήσεων και τέλος ένα ανεξάρτητο ESRTP χρησιμοποιώντας όμως κάποια στοιχεία του VIS και προχωρώντας προς την ενιοποίησή τους. Είναι και η βασική επιλογή μας αν θέλετε. Η πρώτη επιλογή του ανεξάρτητου ESRTP δεν είναι η σωστή επιλογή γιατί δημιουργεί προϋποθέσεις επικαλύψεων. Η δεύτερη επιλογή έχει τους υποστηρικτές της και εδώ αλλά η μελέτη δείχνει ότι παρουσιάζει και αρκετούς κινδύνους. Το να συνδέσει κανείς ένα νέο σύστημα, σε ένα σύστημα λειτουργικό όπως το VIS, λειτουργικό σε 30 χώρες και με απαιτήσει απάντησης 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, θα δημιουργήσει προβλήματα στις οργανώσεις των κρατών μελών. Το πρόβλημα δεν είναι σε κεντρικό επίπεδο, εκεί μπορεί κανείς να προβλέψει τις αλλαγές. Αλλά ε, το πρόβλημα είναι στις επιπτώσεις σε επίπεδο λειτουργίας. Και ένα μάθημα που πήραμε μέχρι τώρα είναι το υψηλό κόστος ε, για τέτοιου είδους λάθη. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Η τρίτη επιλογή την οποία προτιμούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα στοιχεία του VIS, του συστήματος δηλαδή ενημέρωσης Schengen ε, και θεωρούμε ότι είναι και ευθυνότερα από τη δεύτερη επιλογή το συγκεκριμένο σύστημα. Τώρα, ένα επιπλέον στοιχείο είναι η σύνδεση με τα εθνικά συστήματα ES. Είναι μια σημαντική ανησυχία. 13 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν συστήματα συγκρίσιμα με το EES. Αυτά τα κράτη-μέλη για λόγους κόστους και για λόγους οργανωτικούς έχουν ζητήσει τα εθνικά του συστήματα να ενταχθούν πλήρως στο μελλοντικό EES-RTP. Εμείς προτείνουμε να γίνει μέσα από το λεγόμενο National Unique Interface το οποίο θα αναπτύξει με σε κεντρικό τρόπο τα στοιχεία που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση των υπαρχόντων εθνικών ΙΕΣ και ταυτόχρονα ε, θα δώσει ε, στα κράτη-μέλη τα επιπλέον στοιχεία τα οποία δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ε, σήμερα. Δεύτερο σύνολο θεμάτων είναι τα βιομετρικά. Το 2013 στην πρότασή μας εμείς αναφερθήκαμε σαν ε, τον μοναδικό βιομετρικό ε, ταυτοποιητή αν θέλετε ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα. 10 δακτυλικά αποτυπώματα για το ES και 4 δακτυλικά αποτυπώματα για το RTP. Ε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την τεχνική πρόοδο στον τομέα της βιομετρίας και τα πρακτικά προβλήματα καταγραφής υψηλού αριθμού δακτυλικών αποτυπωμάτων στα μεθοριακά σημεία, εμείς προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον αριθμό τους χωρίς να υπονομεύσουμε το σύστημα. Χρησιμοποίησαμε τρεις επιλογές. Μόνο τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα, μόνο φωτογραφία και φωτογραφία προσώπου και τρίτον συνδυασμός δακτυλικών αποτυπωμάτων και ε, φωτογραφίες προσώπου. Ε, βέβαια οι τα καταγεγραμμένα επιπλέον δακτυλικά αποτυπώματα επιτρέπουν τον σωστότερο εντοπισμό και ταυτοποίηση ε, των ε, επιβατών, των ταξιδιωτών. Όταν ενταχθούν στο σύστημα τα βιομετρικά στοιχεία νομίζω ότι μία φωτογραφία ε, ή ένας, ε, ένας φάκελος με δακτυλικά αποτυπώματα θα είναι επαρκής. Θα μας επιτρέψει να κάνουμε ταυτοποιήσεις ε, ταξιδιωτών σε πραγματικό χρόνο στους μεθοριακούς σταθμούς. Έτσι λοιπόν το σύστημα θα γίνει πιο αποτελεσματικό. Και για λόγους ελέγχου και ταυτοποίησης Απαιτείται λοιπόν ένα συνδυασμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων του προσώπου του ταξιδιώτη. Θεωρώντας ότι βασικός στόχος του πακέτου το για τα ευφυή σύνορα είναι η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών σύνορων, η χρήση ε, της φωτογραφίας ως βιομετρικού ταυτοποιητή μόνο ή σε συνδυασμό με ε, έναν περιορισμένο αριθμό δακτυλικών αποτυπωμάτων θεωρείται κάτι το επαρκές και ικανοποιητικό. Βλέποντας λοιπόν το θέμα της βιομετρίας σε επίπεδο κόστους, φαίνεται ότι το σενάριο το οποίο χρησιμοποιεί μόνο τις φωτογραφίες είναι το ευθυνότερο, δεν εκπλήσεται κανείς από αυτό. Υπάρχει μια διαφορά 23 εκατομμυρίων κατέτος σε σχέση ε, με το σύστημα ε, της φωτογραφίας σε συνδυασμό με 10 δακτυλικά αποτυπώματα. Τώρα για τα δεδομένα και την, ε, την κράτηση των δεδομένων αυτών για ένα χρονικό διάστημα. Εμείς είχαμε πει ότι θα πρέπει να κρατάμε τα στοιχεία αυτά για έξι μήνες και για αυτούς οι οποίοι ξεπερνούν τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για 5 χρόνια. Η μελέτη δείχνει ότι μια καλύτερη ευθυγράμμιση αν θέλετε των περιόδων κράτησης των στοιχείων είναι απαραίτητη ανάμεσα στα δύο συστήματα το EES οι έξι μήνες είναι πολύ λίγοι, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσει των διαδικασιών ελέγχου. Αν τα αρχεία των προηγουμένων παραμονών καταργούνται πάρα πολύ γρήγορα, σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να καταγράφονται πολύ πιο συχνά. Σημαίνει επίσης ότι οι μεθοριακοί φρουροί μπορεί να βλέπουν μόνο ένα τμήμα της πρόσφατης μόνον ιστορίας ταξιδιών του συγκεκριμένου πολίτη. Πολλές φορές τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαβατήρια που κρατούν 10 χρόνια, έχουν διάρκεια 10 χρόνων και μπορούν οι μεθοριακοί φορεί να ελέγχουν ε, την προϊστορία, την ταξιδιωτική του συγκεκριμένου ταξιδιώτη με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, λίγο καλύτερα τον χρόνο κράτησης των στοιχείων. Σχετικά τώρα τα λεγόμενα data set Νομίζω ότι μπορούμε να σμικρίνουμε την αρχική πρόταση του ΙΕΣ. E e Είχαμε μιλήσει για 36 στοιχεία. Ο κατάλογος αυτών των στοιχείων μπορεί να είναι και μικρότερος και να φτάσουμε στα 26 αντί για 36. Για το RTP προτείνονται 33 στοιχεία και αυτό δεν αλλάζει. Ένα μικρότερο σύνολο στοιχείων σημαίνει λιγότερος χώρος αρχιοθέτησης και συνεπώς ταχύτερη πρόσβαση στα στοιχεία. Τώρα πάντα στα πλαίσια των δεδομένων θα αναφερθώ λίγο και στη συζήτηση που γίνεται για την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά των αστυνομικών αρχών. Είναι προφανές ότι η μελέτη δεν έχει εξετάσει τα πολιτικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης αλλά έχει ασχοληθεί με το θέμα του κόστους. Ε, θα υπάρχει κόστος για την δυνατότητα έρευνας, αλλά το κόστος αυτό δεν θα είναι πάρα πολύ υψηλό και υπολογίζεται σε 2,5 εκατομμύρια κατέτος. Ε, η διαχείριση γενικά της, του συστήματος δεν αυξάνεται παρά πάρα πολύ λίγο, γύρω στις 200.000 ευρώ το χρόνο. Όταν μπορούν οι αστυνομικές αρχές να χρησιμοποιούν το σύστημα, αυτό μπορούν να το κάνουν αν ε, πράγματι ε, ισχύει τουλάχιστον για έξι μήνες η κράτηση των στοιχείων. Και γι' αυτό ακριβώς, εάν ε, υπάρχει δυνατότητα χρήσης από πλευράς των αστυνομικών αρχών, τότε θα πρέπει να κρατούνται για πέντε χρόνια. Η μελέτη θεωρεί ότι θα κοστίσει 32 εκατομμύρια η επιμήκυνση για την παρακράτηση των στοιχείων αυτών την εποπλέον και αυτό σημαίνει επίσης και 9 εκατομμύρια ευρώ κόστος διαχείρισης το χρόνο. Τώρα, ε, για τις διαδικασίες στις μεθοριακές διαβάσεις. Εμείς εξετάσαμε τα πρακτικά θέματα και τους πρακτικούς περιορισμούς της εφαρμογής των στοιχείων των βιομετρικών στα διάφορα σύνορα. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές ανάλογα όταν έρχεται κανείς με αεροπλάνο, με πλοίο ή με ε, το λοφορείο, με αυτοκίνητα συγγνώμη ή σιδηροδρομικά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας Υπάρχει ένα θέμα χρόνου βέβαια. Μου ζήτησαν να κλείσω την παρουσίαση, γι' αυτό δεν θα περάσω σε επιπλέον λεπτομέρειες. Να πω ότι μία βασική πιθανή λύση θα είναι η λεγόμενη επιταχυντές διαδικασίας. Θα υπάρχει δηλαδή ε, ε, μέσα ε, από περίπτερα να καταγράφονται οι επιβάτες από μόνοι τους πριν φτάσουν στο σημείο ελέγχου κάτι το οποίο θα επιτρέψει τη σμίκρινση ε, της ουράς αναμονής. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πρακτικές λύσεις τις οποίες δεν θα αναφερθώ τώρα. Για τα RTP η μελέτη προτείνει μια διαδικασία εναλλακτική σε σχέση με τα RTP με τις αιτήσει αυτές έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι είναι ήδη καταγεγραμμένοι στο EES να μπορούν online να ζητούν ε, την άδεια εισόδου. Αυτό θα εξοικονομήσει και χρήματα αλλά και χρόνο. Πρέπει να σταματήσω εδώ, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά ελπίζω αν μου κάνετε ερωτήσεις να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Ρόζενμπεργκ. Θέλω να ζητήσω από τους ομιλητές να τηρούν το χρόνο τους παρακαλώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, επόπτη προστασίας δεδομένων, τον κύριο Μπουταρέλη. Έχετε το λόγο κύριε Μπουταρέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να αρχίσω λέγοντας σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε εδώ στη σημερινή αυτή συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το πακέτο ΕΦΗ σύνορα. Είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την πολυπλοκότητα του φακέλου αυτού. Οι προλαλήσαντες ε, σήμερα το απόγευμα αναφέρθηκαν στους στόχους του πακέτου και στην ε, βελτίωσή του. Εγώ κληθήκα εδώ να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στην πτυχή προστασία των δεδομένων και πόσο ξέρουμε ότι μπορεί να ισχύσει στο πακέτο αυτό. Από ό,τι γνωρίζετε, ο προκάτοχός μου είχε εγκρίνει το 2008, το 2011 και το 2015 τρεις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις για το θέμα αυτό. Σε συνεργασία με, 29 ομάδες εργασίας, με την ομάδα εργασίας 29 και με συναδέρφους από τις χώρες μέλη, το 2013 είχαμε μια χωριστή γνωμοδότηση. Η ιδέα του να έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να ελέγχουμε τις εισόδους και τις εξόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι καινούριο. Σήμερα σημειώνουμε την ανάγκη που υπάρχει για νέα βήματα προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την παράτυπη μετανάστευση. Όμως σημειώνουμε επίσης και τις συζητήσεις που γίνονται για την ε, συνεργασία με τις ε, αρχές που ασχολούνται με την μετανάστευση και πώς να εξυγχρονίσουμε τα συστήματά μας. Η προστασία δεδομένων εξακολουθεί πάντως να παίζει ένα σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς ένα σύστημα καταγραφής εισόδων και εξόδων θα οδηγήσει στην επεξεργασία κάποιων πληροφοριών όλων των ατόμων που θα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρόκειται μόνο για τα βιομετρικά στοιχεία. Συνεπώς πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της πρόσβασης στα στοιχεία αυτά των αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό όμω που θέλω να συζητήσω σήμερα με σας είναι να σας πω ότι εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και περιμένουμε, όχι, προχωράμε και εμείς και μελετάμε το θέμα αυτό της προστασίας των δεδομένων και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τον Ευρωπαίο Νομοθέτη να συνεχίζει να εξετάζει την χρήση της τεχνολογίας αφού προηγουμένως έχει καθορίσει συγκεκριμένους στόχους. Είμαστε σε ένα δοκιμαστικό στάδιο σε διάφορα σημεία, σε διάφορες χώρες μέλη, εκεί όπου γίνεται διέλευση των συνόρων. Πώς λειτουργεί αυτό το δοκιμαστικό σύστημα όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα τυχαίνουν ε, επεξεργασίες όσον αφορά τα βιομετρικά στοιχεία, την ίδια και τα δεδομένα του διαβατηρίου. Ποια είναι η νομική βάση Δεν έχουμε αντίρρηση νομικά μιλώντας εφόσον υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία και όλα συνάδουν με τον νόμο και υπάρχει η συγκατάθεση του ατόμου, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από πλευράς προστασίας πάντα δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη συστήματος Λίζα, πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει υποπτή από εμά και από τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Γι' αυτό στην υπηρεσία μας είμαστε σε συνεχείς επαφές με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το σύστημα LISA, LISA ώστε η συλλογή δεδομένων να συνάδει απόλυτα με τις ρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων. Ε, συναντήθηκα πρόσφατα με τον κύριο Γκάρκοφ, τον διευθυντή του συστήματος Λίζα, για να αρχίσουμε να αναλύουμε τις προπτικές που υπάρχουν. Υπάρχει το θέμα των ανώνυμων επίσης δεδομένων. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Εμείς ενθαρρύνουμε όλους τους εκπροσώπους των χωρών μελών να είναι σε επαφή με τους εθνικούς υπόπτες δεδομένων τους για να δουν κατά πόσο διάφοροι στόχοι επιτυγχάνονται ακόμα και σε αυτό το δοκιμαστικό στάδιο χωρίς να κινδυνεύει η προστασία δεδομένων. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα στο μέλλον. Όσον αφορά τη συζήτηση για την ανταλλαγή δεδομένων το PNR, το θέμα είναι ότι πρέπει να τηρείται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα και να τηρούμε βέβαια τις νομικές προϋποθέσεις. Ο κύριος Ντίθ Δεμέρ έχει συμπεριλάβει στην έκθεσή του, στο σχέδιο έκθεσής του, σύσταση όσον αφορά την ανάγκη προστασίας δεδομένων με μία έκθεση αντικτύπου που θα συνεργάζονται οι αρχές προστασίας δεδομένων. Σας ενθαρρύνω λοιπόν όλους σας να διασφαλίσετε ότι η χρήση των επιταχυντών διαδικασίας δεν θα οδηγήσουν σε λιγότερη προστασία δεδομένων. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι για τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε πρωτογενός και δευτερογενός. Τέλος, και αυτή είναι μια άλλη ανησυχία που ακούσαμε και από τον κύριο Κοέγιο σήμερα, είναι ποια τμήματα των συστημάτων που ήδη ισχύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σας ανθαρρύνω λοιπόν να αναλύσετε προσεκτικά τους στόχους και να σκεφτείτε ότι εφόσον εγκριθεί η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναλύεται χωριστά. Πέρα από όλα αυτά, πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά πώς θα εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία, όπου είναι πολύ βασικό στοιχείο το δικαίωμα στην ενημέρωση και να δούμε τι δυνατότητες έχουμε για να τηρήσουμε τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλλαγικότητας. Ένα από τα σχόλια που έκανε ο προκάτοχός μου σχετικά με την γνωμοδότηση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, ο στόχος του μέτρου ήταν σαφής, αλλά το πακέτο τελικά φαίνεται να αρχίζει να ισχύει χωρίς μια σαφή ευρωπαϊκή πολιτική για την διαχείριση των ατόμων που παραμένουν και μετά την λήξη της άδειας παραμονής τους. Φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς έρχονται από χώρες όπου χρειάζεται θεώρηση για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα VIS για να εντοπιστούν. Να λοιπόν ένας ακόμα λόγος για να συνεχίσουμε την ανάλυση και να βελτιώσουμε τη, τους ελέγχους στα σύνορα και την διαχείριση των σύνορων μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να σας ανθαρρύνουμε προκειμένου να χρησιμοποιείτε όπου αυτό δείκνεται τόσα προβλέπει το σύστημα VIS και σας ανθαρρύνουμε επίσης να σκεφτείτε τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα. Εν κατακλείδη, σήμερα εκφράζω την ικανοποίησή μου για την συζήτηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό της προστασίας των δεδομένων και όπως είπα και πριν σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε όλα αυτά τα θέματα και θα είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας για παρετέρω διάλογο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπουταρέλη. Φυσικά. Και υπολογίζουμε όλοι στη δική σας συνδρομή. Τελευταίος ομιλητής τώρα, ο κύριος Γκάρκοφ. Καλωσορίζω τον διευθυντή της υπηρεσίας Λίσα που προβαίνει αυτή τη στιγμή στις δοκιμαστικές εφαρμογές ορισμένων στοιχείων. Θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης του. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Με χαρά είμαστε εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση και η πρωτοβουλία για τα εφή e σύνορα. Υπενθύμησε η Επιτροπή ότι η μελέτη που δημοσιεύθηκε, κατατέθηκε μάλλον πέρυσι, κατέθεσε και μια σειρά συμπερασμάτων και επιλογών. Η πιλωτική δράση της υπηρεσίας μας εφέτος στόχο έχει να προσφέρει περαιτέρω υποστήριξη και τεκμηρίωση στα απέστωρα τα Στοιχεία της εκθέσεως, κυρίως στοιχεία που έχουν να κάνουν με την επιτάχυνση της λειτουργίας των σύνορων και την εμπειρία των ταξιδιωτών στα σύνορα, με την μεταφύση σύνορα. Η πιλωτική η δοκιμαστική αυτή ε, περίοδος δεν έχει στόχο να επαληθεύσει όλα τα στοιχεία. Βεβαίως τα πρωτότυπα έχουν πολύ, μεγάλη σημασία λόγω των τεχνικών επιλογών που εμπεριέχουν και ε, της αξιολόγησης των συνεπειών για τη διαχείριση των συνόρων. Και έτσι λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να συλλέγουμε τις εμπειρίες των συνοριοφυλάκων και των ταξιδευτών που συμμετέχουν στη δοκιμαστική αυτή εφαρμογή. Έχει προσδιοριστεί το πεδίο της δοκιμαστικής εφαρμογής σε συνεργασία στενή με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κρατημέλη. Περιλαμβάνει δε 13, 13 περιπτώσεις δύσκολες με μία σειρά ερωτημάτων, 100 το όλων, που έχουμε εκπονήσει από κοινού με την Επιτροπή, αλλά υπάρχουν και μελέτες επί χάρτου που καλύπτουν αντίστοιχες ε, υποθέσεις που όμως δεν απαιτούν τεχνολογία και τεχνική δοκιμαστική φάση. Τα αποτελέσματα θα κατατεθούν έως το Σεπτέμβριο του 2015 και ως το τέλος του έτους, το Νοέμβριο περίπου, θα έχουμε τελική έκθεση που θα αξιοποιηθεί για τα, για τη διατύπωση συμπερασμάτων στη συζήτηση και την ε, νομοθετική πρόταση που ενδεχομένως θα αναλογιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και την αξιολόγηση προηγούμενης. Για τη σημερινή συζήτηση έχουμε προετοιμάσει τη φάση της δοκιμής, δεύτερη φάση που ξεκινάει το Μάρτιο με 12 κρατημέλη που υποστηρίζουν την ε, δοκιμαστική εφαρμογή και 17 διαφορετικά συνοριακά φυλάκια καθώς μια από τις σημαντικές προθέσεις και αποτελέσματα αυτής της ε, μελέτης είναι να αξιοποιηθούν δοκιμές σε, σε φυλάκια, είτε χερσαία, είτε ε, αεροπορικά, είτε θαλάσσια. Καθίσατε φυσικά σαφές ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαχείριση των συνόρων με την εκτέλεση των πιλωτικών προγραμμάτων εφέτος. Το βλέπουμε ξεκάθαρα και θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι η υπηρεσία μας διαβουλεύτηκε με τον επόπτη προσωπικών δεδομένων στην πρώτη φάση της προσέγγισης και της διαμόρφωσης εκμαστικής εφαρμογής ώστε να υπάρξει πλήρης σεβασμό της ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης η δική μας υπηρεσία δεν πρόκειται να συλλέγει, να ε, αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε όλη αυτή τη φάση. Αυτή τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Εχθές συγκεκριμένα ένα από τα κράτη που συμμετέχουν στη δοκιμαστική εφαρμογή ήρθε και υπέβαλε τις προτάσεις του με βάση και τις αρχές για τη συμμόρφωση στις ε, αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σα διαβεβαιώ λοιπόν ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα υπόψη. Επίση η υπηρεσία μα σχεδιάζει και, εφαρμόζει εκστρατεία ενημέρωση σε όλα τα μεθοριακά φυλάκια, έτσι ώστε όλοι οι ταξιδιώτε να λαμβάνουν την απαραίτητη ενημέρωση και να προσφέρουν τη συνένεσή τους εν ώψη της συμμετοχής τους στη δοκιμαστική εφαρμογή και να αποδέχονται την ενδεχόμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις αρχές των κρατών που συμμετέχουν στη δοκιμαστική εφαρμογή. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι έχουμε και αρκετούς μπλεκόμενους φορείς όπως την υπηρεσία της, των θεμελιωδών ελευθεριών και άλλους φορείς που συμμετέχουν και συμβάλλουν εν τέλει στην τελική έκθεση η οποία θα φωτίσει πιστεύω σε μεγάλο βαθμό και διάφορες τεχνολογικές εναλλακτικές που δοκιμάζονται και τις συνέπειες τους στα θεμελιώδη δικαιώματα. Με αυτήν είναι λοιπόν η δοκιμαστική εφαρμογή καλύπτει όχι μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και συνέπειες τόσο στη διαχείριση των συνόρων όσο και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για να ολοκληρώσω εδώ, έχει ξεκινήσει προετοιμασία σε στενό συντονισμό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εργαζόμαστε, τους ενημερώνουμε τακτικά για την πρόοδο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικό και σημαντικό στοιχείο για μας βέβαια είναι η διαφάνεια και πιστεύουμε ότι χάρη σε αυτήν θα μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάρκοφ και τώρα θα ήθελα να ακούσω τους ομιλητές όσους συναδέλφους θέλουν το λόγο στη συζήτησή μας. Έχουμε 40 λεπτά στη θέσή μας. Έχουμε καταγράψει τους ε, ετούντε το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Άννα Νέμες, επιτρέψτε μου όμως να σας υπενθυμίσω να συμπληρώνετε το ροζ έντυπο ώστε να διευκολυνθούμε στη διαχείριση της συζητήσεως για να έχουμε ως το δυνατόν πιο ουσιαστική και στοχευμένη συζήτηση. Σας καλώ λοιπόν να αξιοποιήσετε την παρουσία των εγκεκριμένων προσκεκλημένων μας. Είμαι δεπεπισμένη ότι με τον διάλογο αυτό που μπορεί να αναπτυχθεί σε πολύ επικοδομητικό πνεύμα διδασκόμαστε ημέν από ό,τι καλό και τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και τους ευρωβουλευτές να λάβουν το λόγο. Και καλό την κυρία Ανανέμες από την Πολωνία, από την οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις τους. Να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Καταρχάς, το θέμα της ευελιξίας του συστήματος στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε. Σήμερα απαιτείται η δημιουργία ενός ικανοποιητικού επίπεδου ασφαλείας στη λειτουργία του συστήματος. Ίσως σε δύο χρόνια τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Απαιτείται ένα σύστημα το οποίο καταρχάς να είναι ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στην ισορροπία η οποία απαιτείται από τη μία στο άνοιγμα το οποίο θα πρέπει να έχει η Ευρώπη και από την άλλη στις ανησυχίες για την ασφάλεια της Ευρώπης διότι δυστυχώς οι απειλές είναι πλέον δεδομένες. Οι απειλές βέβαια δεν είναι οι ίδιες για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη μας την υπάρχουσα κατάσταση. Οι λύσεις λοιπόν θα πρέπει να γίνουν δεκτές από όλους και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί, να βελτιστοποιηθεί και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να είναι φθηνό ή ακριβό. Λέγω ότι θα πρέπει να επιτρέπει τη σωστή λειτουργία των μέτρων και εφαρμογή των μέτρων τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα διότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε σήμερα είναι μια νέα πραγματικότητα, όχι πολύ ευχάριστη και έχουμε θα έλεγα μείνει πίσω. Η σημερινή συζήτηση λοιπόν στην οποία η Πολωνική ΣΕΜΑ παίρνει μέρος ελπίζω να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νέμες. Ο κύριος Όστερμαν. Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία ένα τέτοιο εγχείρημα για τα εφή ε, σύνορα να προχωρήσει και μάλιστα εν ώψη της υποβολής νέας νομοθετικής προτάσεως με προσεκτική ανάλυση και μια δοκιμαστική εφαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών. Έχω λοιπόν μια ερώτηση για τον κύριο Μπέρκοφ. Έχει αποφασιστεί για λόγους κόστους αλλά και χρόνους μόνο κάποια στοιχεία να ε, δοκιμαστούν κάποια στοιχεία του προγράμματος αυτού για τα ευφύη e σύνορα. Ε, πώς αξιολογείτε την επιβάρυνση για ολόκληρη τη διαδικασία τότε. Ευχαριστώ κύριε Όστεμαν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λόπες Αγουιλάρ. Είναι πολύ καλός φίλος της Ρουμανίας ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ από την Ισπανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολιτική παρατήρηση που κάνατε για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που αποκλείονται από το χώρο Σέγγεν παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαιτέρως αυτής εδώ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Εμείς ψηφίσαμε υπέρ της ένταξης της χώρας σας και της Βουλγαρίας στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την διεύρυνση του χώρου Σέγγεν προς την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ αφορά την αρχή εποπτείας για τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη συζήτηση. Κύριε Μπουταρέλη, είναι προφανές ότι εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες σχετικά με το εφικτό ή μη σε οικονομικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλότατα έξοδα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, για την δημιουργία της δεύτερης γενιάς SIS2. Σχετικά τώρα λοιπόν με το SIS, το VIS και όλα αυτά τα τεχνικά θέματα είναι προφανές ότι δημιουργούν ε, υψηλότατα επίπεδα σύγχυσης σε όλους μας και ακόμα και σε μας σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία καθαρά τεχνικής φύσης. Αυτά συζητάμε, αυτά μας αφορούν και ξεχνάμε την πολιτική διάσταση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τα τεχνικά πλεονεκτήματα της κοινή διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. Το θέμα λοιπόν που θέτω αφορά στην συνειδητοποίηση η οποία θα πρέπει να υπάρχει για τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Έχετε κάποιες εμπειρίες. Εσείς συνδέεστε επίσης και με τις εθνικές αρχές εποπτείας προσωπικών δεδομένων. Τι εμπειρίες έχετε, σε ποιο βαθμό ο Ευρωπαίος πολίτης συνειδητοποιεί ε, τα προβλήματα αυτά. Αυτός που θα έρθει να μας επισκεφθεί γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον. Εμείς μας είπατε ότι έχετε σχέση με το Ιουλίζα. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε και φυσικά είναι επίσης δύσκολο να το κατανοήσουν και τα μέλη των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών των κρατών μελών. Τι γίνεται με τους πολίτες λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι λίγο ενήμεροι για αυτά τα οποία γίνονται. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν ε, τι δυνατότητες αμφισβήτησης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρουσιάζονται. Δεν θα έπρεπε να γνωρίσουν τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην καθημερινότητά τους οι εφαρμογές οι νέες για τα βιομετρικά στα πλαίσια του πακέτου εφιών συνόρων. ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι θα προσπαθούν να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα. Λοιπόν, ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται ότι φτάνει στην φάση να περάσει μέσω της διαδικασίας της νομοθετικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταστεί σύντομα ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας προσεκτικά, όχι μόνο εσάς το λέω, αλλά για την επιτροπή σας, για την στήριξη στη χώρα μου. Ελπίζω ότι στο κοκτέιλ αργότερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί σας. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μετατρέψω τη συζήτηση σε συζήτηση για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Εμείς όμως σαν χώρες έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στον τομέα του ελέγχου των συνόρων από το 2010. Παρέχουμε ασφάλεια σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είμαστε τμήμα του πιλωτικού προγράμματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι ανήκουμε στην ευρύτερη ζώνη Σέγγεν και ζητάμε εμείς να κρυφούμε επί της ουσίας και όχι κάθε φορά να μας θέτε θέτεται κινούμενους στους στόχους τους οποίους καλούμεθα να πετύχουμε και βάζετε ένα στόχο τον ένα μήνα, τον επιδιώκουμε να τον πετύχουμε και τον αλλάζετε τον επόμενο. Δεν γίνεται έτσι. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ιταλικής Γερουσίας, ο κύριος Κρίνη. Είναι από το κίνημα των πέντε αστέρων ο κύριος Κρίνη. Λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος πάνω από τρία λεπτά για τον κάθε ομιλητή. Από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την ανάγκη της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, στην οποία αναφέρθηκαν κάποιοι προηγουμένως. Γιατί πρόκειται μπροστά μας ε, για μια πολύ σημαντική πρόκληση, να προσπαθήσουμε δηλαδή να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα σε τεχνολογικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως κάθε φορά που βάζουμε έναν διαφορετικό στόχο, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα πρέπει να βλέπουμε τι συνέπειες υπάρχουν σε επίπεδο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με ποια έννοια το λέγω αυτό. Είπατε λίγο πριν για τη διάρκεια κράτησης των στοιχείων. Σιγά σιγά αυξάνουν οι απαιτήσει για τον έλεγχο, για τη χρήση από τις αστυνομικές αρχές ε, και τα λοιπά, για την επαλήθευση και τα λοιπά. Αυξάνεται και η ανάγκη για την μεγαλύτερη ε, παρουσία των στοιχείων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα επίσης αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων και των υπηρεσιών που θα έχουν ε, πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα αυτό. Και όλα αυτά δεν θα έχουν κάποιο νόημα για την αναγνώριση στοιχείων και προσώπων που έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα ή με την τρομοκρατία, ε, γιατί και οι δύο αυτοί τομείς δεν πρόκειται να είναι τόσο ανόητοι και να παραβιάζουν την παραμονή την οποία έχουν ε, πάρει για μια χώρα και θα σέβονται αυτούς τους ελάχιστους κανόνες. Σε αυτή τη φάση λοιπόν και γι' αυτό το λόγο οι στόχοι μας δεν είναι χρήσιμοι. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε στόχους οι οποίοι να είναι πράγματι χρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Και ο μοναδικός απτός στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι στην ουσία να μέτρα αυτούς οι οποίοι ξεπερνούν το χρόνο παραμονής που τους έχει ε, δοθεί. Αν ο στόχος είναι η απλή καταμέτρηση, τότε ίσως η προσπάθεια την οποία κάνουμε να είναι λίγο υπερβολική, δηλαδή όλα αυτά τα βιομετρικά κτλ. κτλ. Δεν έχει καθοριστεί μια σωστή πολιτική διαχείρισης των προσώπων αυτών που ξεπερνούν τα όρια παραμονής όχι μόνο εντοπισμός, αλλά αυτή στιγμή ε, τυχαία ίσως ανακαλυφθεί ένα τέτοιο πρόσωπο, τι γίνεται, αν έχει ξεπεράσει τον χρόνο, πού βρίσκεται το πρόσωπο αυτό και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχουν ε, πολιτικά ε, στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως να αυξήσει ε, την ταχύτητα επεξεργασίας των στοιχείων, αλλά νομίζω ότι θα επιβαρύνει γενικά τα θέματα αυτά σε επίπεδο ουσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Κοέγιο την Πορτογαλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ρόζενμπερκ για όσα μας είπε. Θέλω να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει ανεβάσει την έκθεση 600 σελίδες. Ε, μπορεί να μην τη διαβάσουν όλοι οι πολίτες, αλλά είναι καλό γιατί ενισχύει τη διαφάνεια. Οπότε συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την ανέβασε την έκθεση αυτή στο διαδίκτυο. Θέλω να επιθυμίσω επίσης και αυτό που είπατε για τη διατήρηση δεδομένων που είπατε ότι για μερικούς λόγους έξι μήνες μπορεί να φτάνουν, αλλά αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου, πέντε χρόνια θα έπρεπε να είναι η διατήρηση αυτή. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και νωρίτερα στην πρώτη συζήτηση, ότι πρέπει να καθορίσουμε με ακρίβεια τον στόχο της προσπάθειάς μας αυτή. Αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε. Και τέλος, κύριε Ρόζεμπερκ εκτίμησε ιδιαίτερα αυτό που είπατε για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είπατε 10 πρέπει να είναι κάτι καλό, γιατί προσφέρει περισσότερη προστασία, αλλά σημαίνει βέβαια και περισσότερες καθυστερήσεις και πιο ακριβώς σύστημα. Ακριβώς όμως γι' αυτό καταλήγω στο πρώτο μου συμπέρασμα, ότι δηλαδή δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να θέλουμε την ασφάλεια με ό,τι κόστος και να είναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα. Δεύτερον, κύριε Ρόζεμπεργκ και κύριε Καρκόφ, δεν έχω τίποτα κατά του δοκιμαστικού προγράμματος, μπορεί να είναι πράγματι πολύ χρήσιμο, η ένστασή μου όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό είναι ότι δεν νομίζω ότι το Ιουλίζα νομικά μπορεί να προχωρήσει. Έχω νομική ένσταση δηλαδή, όχι επί της διαδικασίας. Και μπορεί και να ασφάλω, ίσως. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον φίλο Τιθαμέρα και την ε, κυρία Φαγιόν και τους κοιόδους εισηγητές που συμφώνησαν να ζητήσουν γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας, την οποία και περιμένουμε. Όταν θα την έχουμε, θα ξέρουμε αν έχω δίκιο ή όχι. Πάντως, με τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια συμμερίζομαι την ιδέα που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίποτα δεν θα δεχτεί κάτι που θα μειώνει την ε, θέση του και τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πουταρέλη για αυτά που μας είπε και για την επιμονή του όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Κύριε Πουταρέλη, είμαστε κάτι σαν το watchdog όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και την προστασία των δεδομένων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Οπότε, να τηρείτε το χρόνο σας. Δύο λεπτό καθένας. Ο συνάδελφός μας από την Πορτογαλία. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χωζέ Μανταχάλας, ευρωβουλευτής από την ομάδα των σοσιαλιστών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η Πορτογαλία έχει ήδη καταγράψει θετική εμπειρία. Εγκαίρως προχώρησε στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού διαβατηρίου. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια πολιτών που ζήτησαν το ηλεκτρονικό διαβατήριο πέρυσι. Και άλλα κράτη υποστηρίζουν την ε, εισαγωγή του συστήματος φερειπίν τα πορτογαλόφωνα κράτη της Αφρικής που θεωρούν ότι είναι καλύτερη, καλύτερο το σύστημα με το ηλεκτρονικό διαβατήριο. Έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί ικανοποιητικά και με γερές τεχνικές βάσεις λοιπόν. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο δείχνει ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια για να βρούμε μια πραγματικά αποτελεσματική λύση. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συστήματα και σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχει πει ο Επίτροπος ότι η αδράνεια δεν είναι λύση. Δεν έχουμε περιθώριο να μείνουμε αδρανείς και πιστεύω θα πρέπει να αναλάβουμε δράση στα σύνορα, ειδικά εκεί που σημειώνονται περισσότεροι κίνδυνοι. Υπάρχουν σημεία με ενισχυμένους ελέγχους που δεν αρκούν όμως, γιατί αν κάποιος ξεπεράσει το χρόνο παραμονής του ή αν αγοράσει, όπως συμβαίνει καμιά φορά για λόγους ε, ε, οργανωμένου εγκλήματος τη θεώρηση του διαβατηρίου, αυτοί δεν, αυτές οι περιπτώσεις δεν καλύπτονται. Και έτσι πιστεύω ότι η τεχνολογία μόνο δεν αρκεί Μερικέ φορέ δίνεται η εντύπωση εδώ στο Κοινοβούλιο ότι μόνο με, με τα τεχνολογικά μέσα λύνουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ τον κύριο Ρόζενμπορκ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώ μπορεί να βρεθεί μια συμβαστική ε, διέξοδο, μια συμβαστική λύση. Εγώ διρωτώ με εάν υπάρχει δυνατότητα για ένα απλοποιημένο σύστημα μια πλατφόρμα θα έλεγα συνεργασίας μεταξύ εκείνων που ήδη έχουν ένα σύστημα εφιών συνόρων και εκείνων που θέλουν να εισαγάγουν ένα, ένα τέτοιο σύστημα. Μια πλατφόρμα η οποία θα επέτρεπε τη συλλογή των πληροφοριών και την διάθεσή του στα εμπλεκόμενα κράτη. Αυτό είναι μια ερώτηση για τον κύριο Ρόζενμπορ, αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Η δε προστασία των προσωπικών δεδομένων για τον κύριο Μπουταρέλη. Δεν έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν ισχύει αυτό για όλους μας. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ τουλάχιστον να έχουμε μια συνενετική λύση και τα κράτη να, αποτρε... αποφεύγουν κινήσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη καθυστέρηση την εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος. Η τρομοκρατία ως απειλή είναι πραγματική, πρέπει να τη δούμε, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και εμείς στο κοινοβούλιο μας, στο κοινοβούλιο της ε, Πορτογαλίας, σκοπεύουμε να αναλάβουμε πιο σκληρά ακόμα μέτρα κατά των τσιχαντιστών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μια ερώτηση που ακούστηκε από πολλούς ομιλητές, εάν το πακέτο για τα εφή e σύνορα, οι προτάσεις για τα εφή e σύνορα μπορούν να ενισχύσουν το επίπεδο ασφάλειας για τον πολίτη. Και αν μπορούμε να έχουμε αυτό το χώρο της ελευθερίας διακίνησης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, χάρη στα εφή e σύνορα. Μια ερώτηση προς όλους, μια ερώτηση που ακούστηκε από πολλούς. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Και τώρα με τον εκπρόσωπο του και Κέμψη Λίμπερκ, παρακαλώ, και σας καλώ όλους να περιορίσετε τις ομιλίες σας στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, τα στοιχεία εισόδων-εξόδων ε, υπηκών των ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκών τρίτων κρατών, περί τα 600 εκατομμύρια με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα διατήρησης τέτοιου υψηλού αριθμού δεδομένων. Ο κύριος Βοταρέλη, αν κατάλαβα καλά, μας λέει ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα επέτρεπε αν ο πολίτης ή του κράτους ε, που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την άδειά του, να καταγράφονται τα δεδομένα αυτά. Και ρωτώ, θέτω μάλλον το ζήτημα, διότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και κυρίως το Μαυροβούνιο Θα ήθελα να ρωτήσω αν λογιζόμαστε ως τρίτες χώρες ή όχι. Είμαστε χώρες που έχουμε συνάψει συμβάσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι από το Μαυροβούνιο αν ταξιδέψουμε είτε προς τις μας είτε προς Ανατολά από τα 20 μέχρι τα 100 χιλιόμετρα απόσταση βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κροατία είναι αυτή, Ιταλία είναι αυτή, Ελλάδα είναι αυτή. Άρα λοιπόν το λέω διότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ως προς την εφαρμογή του πλαισίου εφιών συνόρων για τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Winberg, Σουηδία παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει και το θέμα των χρυσών θεωρήσεων, οι οποίες προβλέπονται για να αποφύγουν την αναμονή. Αυτοί που θα ζητήσουν όμως αυτές τις θεωρήσεις, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Ε, και φυσικά ανάμεσα στους πλουσίους υπάρχουν και τρομοκράτες. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξή. Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα ελέγξετε αυτού του τύπου τα πρόσωπα. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να του ελέγξετε αυτή τη στιγμή επιστρέψουν από, τις, από τα διάφορα ταξίδια τους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τρομοκράτες μπορεί να εισχωρήσουν στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών εύκολα και δεν κάθονται να περιμένουν ουρά Λοιπόν καλό είναι τα ευφυή σύνορα, αλλά καλύτερη είναι η ασφάλεια των σύνορων και στη συνέχεια να δούμε τι θα κάνουμε με την ευφυΐα των σύνορων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί λίγο καλύτερα τα συστήματα που έχει ε, στην διάθεσή της σήμερα. Το Eurodact ε, δεν λειτουργεί και πολύ. Το Frontex λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Mare Nostrum ε, το σύστημα και εκεί δεν ήταν πολύ ικανοποιητικό. Γι' αυτό λοιπόν αντί να φτιάχνετε καινούργια φτιάξτε τα παλιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο. Στον εκπρόσωπο του Τουρκικού Κοινοβουλίου. Στον κύριο Ντίνκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. οι ελευθερίες και η δημοκρατία πρέπει να βρίσκονται σε ισότιμο επίπεδο μέσα στα δημοκρατικά κράτη. Αν ανατραπεί αυτή η ισορροπία δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία. Και για τη θεώρηση και στα υπόλοιπα θέματα ε, που συζητούμε μέσα στο πλαίσιο των ευφυών συνόρων πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αρχές της ελευθερίας και την ασφάλεια σε μια ισορροπημένη σχέση. Το σύστημα πληροφοριών ε, Schengen αναφέρεται και στη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με ένα σύστημα πληροφοριών βράχυπρόθεσμων προσωπικών στοιχείων για τη θεώρηση των διαβατήριων. Ένα σύστημα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστημα αξιόπιστο, τα χρησιμοποιεί και η Τουρκία, και έχουμε τους ε, υπηκόους οι οποίοι καταθέτουν την αίτησή τους, δίνουν δακτυλικό αποτύπωμα και φωτογραφία και ως εκ τούτου έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο σύστημα θεωρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από κράτη άλλα κράτη, εκτός αυτού που τα καταγράφει, εφόσον ε, διατυπωθεί το σχετικό αίτημα, ή να διορθωθούν αναλόγως αν υπάρχουν εσφάλματα. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά, λοιπόν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ζήτημα της ε, κοινή χρήσης των δεδομένων και στο θέμα της θεώρηση των διαβατηρίων, θα ήθελα να παρακαλέσω, κυρία Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων για του υπηκού Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ζήτημα το οποίο συζητούμε εδώ και καιρό και που περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε ένα νοδικό χάρτη με συγκεκριμένα ε, στάδια τα οποία έχουμε υλοποιήσει. Με την έκθεσή της στις 20 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιβεβαίωσε άλλωστε και έχουμε αναπτύξει, σημαντικό νομοθετικό αλλά και τεχνολογικό πλαίσιο ώστε να ικανοποιήσουμε τους όρους για την απαλλαγή από τη θεώρηση διαβατηρίου. Περιμένουμε χρόνια για να υλοποιηθεί αυτή η προσδοκία μας. Έχουμε κάνει το μερίδιο από πλευράς μας της δουλειάς και περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο θα λάβει ο συνάδελφος από την Κροατία, Νενάτ Σταζίκ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Hrvatska nije dio Schengena e, i nadamo se da ćemo to postati što je moguće prije, ali to nije tema ε, Κυρία Πρόεδρε, η Κροατία ανοίξει το χώρο του Σέγγεν. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να, να δημιουργήσει προβλήματα. Φυσικά το νέο σύστημα θα έχει κόστος, θέλουμε να είναι αποτελεσματικό, θέλουμε να είναι αναλογικός προς τη δαπάνη και να εξασφαλίζει βέβαια την ε, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 200 εκατομμύρια υπηκόους τρίτων κρατών, για τους οποίους μπορεί να έχει ακόμη και αποτρεπτικό χαρακτήρα ένα τέτοιο νέο σύστημα, διότι ε, δεν προτιμά κανένας πολίτης να χορηγεί βιομετρικά στοιχεία, ειδικά αν πρόκειται αυτά να αποθηκευθούν για έξι ή και περισσότερους μήνες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορεί να, έχουν, ε, μπορεί να τρέφουν φόβους για το πώς θα αξιοποιηθούν ε, αυτά τα στοιχεία οι πολίτες. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει το εξής. Εάν είναι λόγος ανάπτυξης επιφυλακτικότητας και δεχομένως να έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα το νέο αυτό σύστημα αποτρεπτικό θα έλεγα για υποψήφιους τρομοκράτες, τότε ναι, αλλά δεν θα ήθελα να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα για τους πολίτες, τους φιλιρινικούς πολίτες των κρατών που θα ήθελαν να επισκεφθούν χώρες δικές μας και βέβαια αυτό θα επηρεάζει όπως καταλαβαίνετε σημαντικά τον τουρισμό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντίαθ Ντεμέρα. Είναι ένας από τους εισηγητές μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μια γενική ερώτηση πρώτα. Γιατί δεν έχουμε όλη την υποχρέωση να τα ξέρουμε όλα. Και εγώ, πρώτος και καλύτερος, μαθαίνω πολλά και ξέρω ότι κάθε λεπτό της ζωής μου έχω να μάθω πολλά. Και σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, ο κανόνας. Ακόμα δεν υπάρχει, δεν έχουμε τον κανόνα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι κάνουμε υποθέσεις για έναν κανόνα που ήδη υπάρχει στα χαρτιά, αλλά που θα τροποποιηθεί, όπως είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος. Άρα δεν υπάρχει. Επιπλέον πρέπει να προσθέσω ότι η προστασία δεδομένων είναι κύριο δικαίωμα, Φερνάντο. Κύριο. Και κάθε κανονισμός ή κάθε οδηγία πρέπει να τηρεί αυτό το πρωτογενές δίκαιο, το κύριο δίκαιο. Συνεπώς, εντάξει, όταν θα έχουμε ό,τι στοιχεία χρειαζόμαστε, με τη βοήθεια των Εθνικών Κοινοβουλίων βέβαια, τότε θα ετοιμάσουμε το κανόνα. Και κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας θα αποφασίσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε σε οποιαδήποτε παρέκβαση από το κύριο αυτό δίκαιο. Κύριε Ρόζενμπουργκ, σας ευχαριστώ. Αυτό μόνο έχω να σας πω σήμερα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε πάντα στη διάθεσή μας για να έρθετε και να μας τα εξηγήσετε. Γιατί, εντάξει, και εγώ τα είπα όλα αυτά από την τεχνική έκθεση, τις διάφορες επιλογές, α, β, γ κτλ. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ε, κοινή, μη κοινή, αναγνώριση προσώπου ή όχι. Ωραία. Καλά προχωράμε. Προς τον κύριο Καρκόφ όμως. Το ίδιο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει η Τάνιο και εγώ μαζί σας ήταν πριν από δύο ώρες. Για το δοκιμαστικό πρόγραμμα και το πώς θα εξελιχθεί και για την προστασία δεδομένων. Πάλι κύριο δικαίωμα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περίοδου. Αυτός με τον οποίο δεν μιλήσαμε τόσο, όχι γιατί δεν ήθελα αλλά γιατί δεν είχαμε χρόνο, είναι ο κύριος Μπουταρέλη. Ο κύριος Μπουταρέλη είναι πολύ βασικός στην προστασία δεδομένων. Ανέλαβε τα καθήκοντά του βέβαια πρόσφατα ως νούμερο ένα, αλλά έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό που ασχολείται με την προστασία των δεδομένων. Για μας λοιπόν αποτελεί εγγύηση αυτό. Θέλω λοιπόν σε αυτό να απευθύνω μία από τις αμφιβολίες μου. Είπατε ότι δοκιμαστική περίοδος, κατά την ε, περίοδο αυτή δηλαδή, οι εθνικοί επόπτες ε, και οι πρόσωποι του θα φροντίσουν για την προστασία των δεδομένων. Εξηγήστε το μου αυτό καλύτερα. Στην περίπτωση που, υποθετικά το λέω έτσι, που οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν πρόσβαση στο νομοθετικό πακέτο. Είπατε κύριε Μπουταρέλη, διαφορετική μεταχείριση και χρησιμοποίησατε τον όρο αναλογικότητα που πολύ μου αρέσει εμένα. Αναπτύξτε μου σας παρακαλώ αυτές τις έννοιες στην περίπτωση που οι αρχές επιβολής του νόμου θα είχαν πρόσβαση. Τίποτα άλλο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε δύο κυρίες από τα Βαλκάνια που προεδρεύουν τις σημερινές μας συνεδριάσεις. σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία δίχως άλλο να συζητήσουμε παρετέρω τα σημερινά θέματα και αργότερα στη δεξίωση που θα ακολουθήσει μετά την συνεδρίαση αυτή. Προηγουμένως όμως θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν. Ε, εγώ θα κακιά τώρα, γιατί πρέπει να σας ζητήσω να περιοριστείτε σε τρία λεπτά. Κύριε Ρόζεμπερ πρώτα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την ερώτησή σας. Το σύστημα αυτό θα παρέχει την ασφάλεια που επιθυμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και η ερώτηση χρειαζόμαστε ασφαλή σύνορα ή ευφυή σύνορα. Κοιτάξτε, στόχος μας είναι τα ευφυή σύνορα να είναι και πιο ασφαλή. Ταυτίζεται αυτό. Όπως εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο μεθοριακός φουρός όταν ελέγχει έναν εκπρόσωπο τρίτης χώρας ε, εξετάζει πολλά πράγματα. Ελέγχει το ταξιδιωτικό έγγραφο ελέγχει λοιπόν την αυθεντικότητά του, αν του ανήκει. Θα πρέπει να ελέγξει επίσης αν έχει μια θεώρηση εφόσον απαιτείται. Θα πρέπει να δει αν υπάρχει μια προειδοποίηση για το πρόσωπο αυτό στα πλαίσια του VIS και θα πρέπει να ελέγξει επίσης και το αν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει σεβαστεί ή μη μια προηγούμενη παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνώντας ε, την παραμονή αυτή, κάτι το οποίο οδηγεί σε απαγόρευση εισόδου. Όλα αυτά πρέπει να τα ελέγξει ο τέλος συνοριακός φορός, αυτό είναι δύσκολο και χρονοβόρο και υπάρχει και έλλειψη μέσων κτλ. Λοιπόν, το σύστημα είναι να βοηθήσουμε τον ε, μεθοριακό φρουρό να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τεχνολογία. Το θέμα δεν είναι στατιστικό μόνο. Προφανώς πρέπει να τροφοδοτηθούν και οι στατιστικές. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στο μεθοριακό φρουρό να κάνει τη δουλειά του σωστά σύμφωνα με τον κώδικα του Σέγγεν. Δεύτερον, Ε, μπορούμε να φτιάξουμε μια μικρότερη πλατφόρμα για τη συμμετοχή των κρατών μελών. Εδώ η απάντηση είναι ότι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το βλέπει. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σύστημα απλούστερο από αυτό που είχε προταθεί, ευθυνότερο, αποδοτικότερο, πιο ελαφρύ γραφειοκρατικά και για τους μεθοδιακούς σκοπούς και για τις προξενικές αρχές, ένα ταχύτερο σύστημα και όπως είπα να κοστίζει λιγότερο. Και γι' αυτό η πρότασή μας είναι και πιο ευφυής θα έλεγα από αυτήν που παρουσιάσαμε το 2013. Πάντα στα πλαίσια του συστήματος Schengen αλλά ταχύτερο και ευθυνότερο κάτι το οποίο είναι καλό και για τον τουρισμό, γιατί θα πρέπει να επηρεάσουμε θετικά τον τουρισμό, δεν θα πρέπει ε, να παρεμποδίζουμε την είσοδο των τουριστών, πρέπει να τους επιτρέπουμε ταχύτερη είσοδο. Τώρα για τον κύριο Κουέλιο σχετικά με την κράτηση την χρονικά πέντε χρόνια για τις αστυνομικές αρχές. Αυτό είναι το λεγόμενο επίπεδο στάνταρντ όπως ισχύει. Υπάρχει και στα πλαίσια του VIS το αντίστοιχο. Ε, σε κάποιες χώρες ε, και για το Eurodac είναι πέραν των 5 ετών. Αλλά η μελέτη προτείνει και το είπαμε και το 2013 ότι αν υπάρξει πρόσβαση των αστυνομικών αρχών στα στοιχεία αυτά πρέπει να κρατούνται τα στοιχεία 5 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που βολεύει και τους ίδιους τους ταξιδιώτες νομίζω. Όπως εξήγησα ήδη ότι αν δεν υπάρχουν ε, πληροφορίες για τον ταξιδιώτη σε ένα σύστημα αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά πρέπει να επανεγγράφεται. Αυτό σημαίνει ότι ξεχνάμε ε, είναι κάτι το οποίο βοηθάει τους ίδιους τους ταξιδιώτες οι οποίοι θα μπορούν ταχύτερα, ταχύτερα να περνούν από τα σημεία ελέγχου και αυτό θα βοηθά επίσης και τους μεθοριακούς σκοπούς ε, να ελέγχουν ταχύτερα. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε τη διάσταση αυτή. Υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δέκα δακτυλικά. Ναι, δεν χρειάζονται δέκα δακτυλικά, αυτό το είπαμε. Εγώ νομίζω ότι θα προτείνουμε και θα περάσει η νέα πρόταση, δεν θα υπάρχουν δέκα δακτυλικά εκεί αυτό που είπα ότι ο συνδυασμός της φωτογραφίας και των τεσσάρων δακτυλικών είναι θα έλεγα ε, το ίδιο επίπεδο ασφαλείας ε, από ότι τα δέκα δακτυλικά είναι ταχύτερο και εφαρμόζεται πιο εύκολα. Αν δεχθεί κανείς λοιπόν ένα χαμηλότερο ε, επίπεδο ασφαλείας μπορεί κανείς ε, να μειώσει ακόμα περισσότερο τα δακτυλικά ή και να τα καταργήσει πλήρως. Και σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ντεμέρα συνεχίζουμε την συζήτηση, συναντώμεθα τακτικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όταν λοιπόν ε, υπάρξει η τελική πρόταση θα πρέπει σε τεχνικό επίπεδο να βρεθούν λύσεις σε όλα αυτά τα επιμέρους θέματα. Γι' αυτό έγινε αυτή η σημαντική μελέτη και ελπίζω να μπορέσουμε να περάσουμε στην φάση ελέγχου, στο test phase. Και ένα τελευταίο σημείο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, αναγκαιότητα, αναλογικότητα. Αυτά είναι θέματα που τέθηκαν από τον κύριο Μπουταρέλη να είστε σίγουρος ότι αυτό ισχύει και για μας. Το σεβαστήκαμε και στην πρόταση του 13 και εξακολουθούμε να το σεβόμεθα και σήμερα. Και είχαμε μία σειρά ανταλλαγών απόψεων με τα κράτη-μέλη και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ότι πράγματι η πρόσβαση στα στοιχεία των αστυνομικών δυνάμεων γίνεται με σωστό τρόπο θελήσαμε να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο συστήματος Σέγγεν και σε επίπεδο ε, συστημάτων αυστηρά εθνικών. Τα ευρήματά μας ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως μπορώ να πω από την πρώτη φάση και γι' αυτό δεν έχουμε πιστεί ακόμα απολύτως ότι είναι αναλογικά απαραίτητη η πρόσβαση των αστυνομικών αρχών. Ο κύριος Μπουταρέλη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για τις ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν. Από την ε, Πολωνή βουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, ευελιξία και ανοιχτή προσέγγιση με προσανατολισμό στο μέλλον βεβαίως δεν, αποκλείεται, δεν αποκλείουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφόσον όμως είναι απόλυτος εξασφαλισμένη η τήρηση των κανόνων Πρέπει να, είμαστε, πρέπει να υπάρχει και η έννοια της ισονομίας ως προς την ε, ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τον κύριο Λόπες Αγγελάρ, η ερώτησή σας ως προς την ε, ευαισθητοποίηση. και πόσο είναι δεδομένη η ιδέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πόσο είναι σημαντική για το μέσο πολίτη. Κοιτάξτε, είναι... Θα ήταν πρόχειρο να κάνουμε μια αξιολόγηση μόνο με βάση τις ανάγκες. Ε, με τις τεχνολογικές λεπτομέρειες και τις ε, και τεχνικά χαρακτηριστικά αξιολογούμε ένα σύστημα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει βεβαίω η δυνατότητα ένα σύστημα εισόδων-εξόδων το οποίο να προσφέρει προσθεμένη αξία στις αρχές μετανάστευσης. Αλλά τι, τι θα πούμε για την ε, ενισχυμένη παρέμβαση στα προσωπικά δεδομένα. Μην θεωρείτε λοιπόν ότι ε, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι απλώς μια σύσταση. Το δικαστήριο ορίζει όρους, προϋποθέσεις και εγώ θέλω να σας βοηθήσω βεβαίως στην αξιολόγηση αυτών των ε, αναγκών αλλά σας παρακαλώ και να λάβετε υπόψη πως σε περίπτωση αμφισβητούμενης αναγκαιότητας το ίδιο μέτρο θα είναι εξίσου αμφισβητούμενο για τον κύριο Πρίμη επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην απάντησή μου με μια από τις τρεις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τρεις πιο διαδεδομένες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπω να διαβάζετε μια ανακοίνωση που αναφέρεται και σε μια δική μας τοποθέτηση για τους ε, ταξιδιώτες βραχίας παραμονής που δεν είναι ύποπτοι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, γιατί φαίνεται ότι το παλαιότερο σύστημα, είπε ο κύριο Δεμέρα, ότι περιμένουμε, ότι περιμένουμε την ε, νέα πρόταση. Με την παλαιότερη όμως τι συνέπεια θα είχε η παλαιότερη για όποιον ε, υπερεύαινε τα όρια της θεώρησης, τα χρονικά όρια, ε, θα ήταν ίσω αδυνατό να λάβει νέα θεώρηση ή Φερρυπίν θα μπορούσε ο εντοπισμός κάποιου που έχει ξεπεράσει τα χρονικά όρια να βοηθούσε στην ε, ενίσχυσή του στην επάνωδο στην πατρίδα του. Αλλά με το νέο σύστημα τι περισσότερο μπορούμε να προσφέρουμε για τον Πορτογάλο συνάδελφο και εκτιμένον ναι, πρωτογενές δίκαιο βεβαίως, άρα δεν υπάρχει εμβολία ότι θα στηριχθούμε πάνω σε αυτό. Για το Μαυροβούνιο και την ερώτησή του, η συνένεση δεν θα ζητείται ανάλογα με την υπηκότητα του ερωτωμένου. Θα ισχύει για τους πάντες ή για κανέναν. Το ζήτημα είναι εάν το σύστημα στη χώρα σας επιτρέπει την επεξεργασία επιπλέον πληροφοριών. Η προτελευταία ερώτηση για τη Σουηδία, για το αν τα εφή e σύνορα θα πρέπει να εισαγάγουν ε, νέα συστήματα. Δεν βλέπουμε εδώ τίποτε το ουσιαστικό. Σε σχέση με το τι κάνουν τελικά αυτοί που ξεπερνούν τα χρονικά όρια της θεωρησής τους. Απλώς έχουμε ένα σύστημα που καταγράφει θετικές ή αρνητικές ε, παρατηρήσεις. Παρέμεινε περισσότερο ή όχι. Για τον κύριο Διεσδεμέρα επίσης. Εξετάζουμε τώρα τις προϋποθέσεις για την εκκίνηση ενός πιλωτικού προγράμματος η Λίζα μας λέει ότι θέλει να καταγράφει, να επεξεργάζεται πλήρως ανώνυμες πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει χωριστή πρόσβαση στη δοκιμαστική εφαρμογή για τις αρχές επιβολής του νόμου. Κύριο Σκάρκοφ και ευχαριστώ πολύ που θα περιοριστείτε στα τρία λεπτά απολύτως. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ έτσι κι αλλιώ θα αλλάξουν τα πράγματα ε, μετά τα συμπεράσματα της δοκιμαστικής περίοδου. Να απαντήσω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα για το πεδίο εφαρμογής. Είμαι προηγουμένως να υπενθυμίσω ότι τώρα βασιζόμαστε σε απόφαση που είχαν πάρει παλιότερα οι χώρες μέλη. Οπότε από πλευράς των χώρων μελών είχαμε τον καλύτερο συμβιβασμό του να τηρούνται τα περιθώρια και των άλλων υποχρεώσεων που είχαμε. Πρέπει εδώ να τονίσω πάντως ότι το δοκιμαστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και διάφορα στοιχεία τα οποία μας φέρνουν ε, πιο κοντά στο πιο επιθυμητό σενάριο από τις χώρες μέλη. Είμαι πεπισμένος ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και για να βοηθήσουμε όσους αποφασίζουν. Η υπηρεσία μας συνεργάζεται πάντως στενά με τις χώρες μέλη, που πολλές φορές όπως η Φιλανδία και η Γερμανία έχουν αντίστοιχες προσπάθειες. Μετά από μερικούς μήνες θα μπορούμε να ανταλλάξουμε λοιπόν απόψεις, έτσι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει ακόμα περισσότερο νόημα. Τώρα, κατά πόσο προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και προστασία στους πολίτες ένα τέτοιο σύστημα, η απάντησή μου είναι ότι δυνητικά ναι. Αλλά μέσα στους επόμενους μήνες όλοι πρέπει να κάνουμε κάποιες ευφύς επιλογές που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική του συστήματος, αλλά θα πρέπει να διδαχτούμε από το παρελθόν να κοιτάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν εναρμονισμένα τα τεχνολογικά μέσα. Γιατί είναι χρήσιμα εφόσον χρησιμοποιούνται και πλήρως. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την τεχνολογική διάσταση. Εν κατακλείδη πιστεύω ότι όντως τεθεί σύνορα μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ε, πρόσθετη αξία που προσφέρουν τελικά στον Ευρωπαίο πολίτη και από τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές μας. Επιτρέψτε μου επίσης να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Και τέλος ευχαριστώ την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την γραμματεία της Επιτροπής αυτής και όσους είναι υπεύθυνοι για τη σχέση μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά να, μια ευκαιρία για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας άτυπα είναι στη δεξίωση που λαμβάνει η χώρα τώρα έξω από την αίθουσα. Αύριο το πρωί στι 9 θα τα ξαναπούμε στην ίδια αίθουσα. Και πάλι καλό βράδυ.